του Αλγερίου καθώς και την ατζέντα του Σαχέλ. Θα περιοριστώ σε μια γενική παρουσίαση, να σας φτιάξω ένα δηλαδή συνολικό πίνακα της ε, κατάστασης. Όσον αφορά την κατάσταση θα πρέπει να έχει κανείς υπόψη του όταν ενδιαφέρεται για τη ζώνη Σαχέλ ότι είναι μια περιοχή κοντά στην Ευρώπη και όπου κάθε συνιστόσα της ε, και βεβαίως εκεί τίθεται και θέματα μετανάστευσης και πρόκειται για μια, πραγματικό, μια ε, τεράστια ζώνη που μπορεί να θεωρηθεί στρατηγική και που περιλαμβάνει την Ευρώπη, την Βόρεια Αφρική και την ίδια την Σαχέλ. Και τα χαρακτηριστικά της δεν είναι πολύ διαρθρωμένα. Βλέπει κανείς και τη μεγάλη δυσκολία της κατάστασης που αντιμετωπίζουμε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει καθορίσει την Σαχέλ μέσα από τη στρατηγική για το Μαλί, την Μπουρκίνα Φάσο, το Τσάτ κλπ. Πέντε χώρες συνολικά για την κατάσταση της ΑΕΛ και είναι ένα μεγάλο μέρος ωστόσο και των χωρών της ε, Βόρειας Αφρικής και της Δυτικής Αφρικής που έχουν και άμεσες διασυνδέσεις με την Ευρωπαϊκή Ήπειρο και αυτό είναι το μέγα χαρακτηριστικό της κατάστασης αυτής της ΑΕΛ ότι είναι μια τεράστια ζώνη και η οποία μάλιστα προσεγγίζει την Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Έχουν γίνει πρόοδοι τα τελευταία χρόνια η στρατηγική για τη Σαχέλ χρονολογείται εδώ και τέσσερα χρόνια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες χώρες συμμετέχουν, κάτι που δείχνει το ενδιαφέρον της διεθνούς κοινότητος για την ζώνη Σαχέλ. Ένας αριθμός λοιπόν βημάτων πρόοδου έχουν γίνει στο στρατιωτικό επίπεδο, ιδίω χάρη στην ε, γαλλική παρέμβαση, ιδίω στο Μαλί, μετά όμως προχώρησε στην περιφέρεια γενικότερο μετά από την παρέμβαση Μπαρκάν τον Νίγηρα που είναι στο επίκεντρο των ε, εξελίξεων αυτών και το στο Μαλί, το Μπόκο και ούτω καθεξής. Και επομένως πρώτα μια σταθεροποίηση στρατιωτική χάρη στην διεθνή παρέμβαση που έχει και μια ουσιώδη συνιστόσα, μινουσπάν δηλαδή την ε, δύναμη των Ηνωμένων Εθνών στο Μαλί υπάρχει και μια θέληση οργάνωσης των χωρών αυτών σε αυτό που ονομάζουν G5, να προχωρήσουν δηλαδή σε μια κοινή περιφερειακή οργάνωση και συνεργασία μέσα σε μια κατάσταση που βεβαίως έχει περιφερειακό χαρακτήρα με πολλές διασυνδέσεις που και αυτές δεν είναι διαρθρωμένες μεταξύ των διαφόρων αυτών χωρών της ε, περιφέρειας. Άλλη σημαντική θετική εξέλιξη ήταν οι συνομιλίες, βλέπετε η συμφωνία της Ουαγκαντούγκου για τη σταθεροποίηση του Μαλή εδώ και δύο χρόνια που είχε ως στόχο να επιτρέψει τη εξαγωγή εκλογών στο Μαλή και τώρα τις συζητήσεις του Αλγερίου που οδήγησαν σε μια συμφωνία η οποία σε στάδια, ελπίζουμε βέβαια, θα μπορέσει να υπογραφεί από το σύνολο των πρωταγωνιστών το επόμενο Σάββατο στην Μπαμακό. Και θα ήθελα να προσθέσω επίσης ότι πίσω από αυτά ή γύρω από όλα αυτά γίνονται και προσπάθειες για να ε, γίνει μια συμβολή σε μια σταθερότητα πολιτική σε όλες τις χώρες αυτές και στο Μαλί μετά το πραξικοπήμα και στην Πουρκίνα Φάσο που είχε κάποιες ταραχές πέρσι και που σήμερα βρίσκεται σε μια διαδικασία σταθεροποίησης η οποία εξελίσσεται καλά. Αυτά βέβαια είναι θετικές παράμετροι που δείχνουν ότι με την όθηση και την υποστήριξη της διεθνούς κοινότητας μπορούν να απτυχθούν κάποιες θετικές δυναμικές. Βέβαια είναι σαφές ότι η ανασφάλεια επί τόπου εξακολουθεί να είναι σημαντική και μάλιστα η τάση της είναι να μεγαλώνει, παράδειγμα Μπόκο Χαράμ, παράδειγμα η κατάσταση στη Λιβύη. Η κατάσταση στο Μαλί επίσης είναι πολύ εύθροστη, υπάρχουν τρομοκρατικές ομάδες οι οποίες έχουν αποδυναμωθεί Άλλες όμως παραμένουν αρκετά ισχυρές και υπάρχει και τάση επέκταση του φαινομένου αυτού. Νομίζω ότι γνωρίζετε για τις απόπειρες που έγιναν σήμερα το πρωί στο Τσάντ και που δείχνουν την αύξηση της επιρροής των ομάδων αυτών, καθώς επίσης και απόπειρες στο νότο του Μαλή πριν από λίγες μέρες. Δεν είναι πολύ καθαρό πάντοτε ποιος κάνει τι. Όμως η ζώνη ανασφάλειας διευρύνεται. Από την άλλη μεριά μπορεί να πει κανείς και ότι όλες οι διεθνείς προσπάθειες δεν έχουν τροποποιήσει τις βασικές παραμέτρους της καταστάσεως, δηλαδή την ευθραστότητα των κρατών, των κυβερνήσεων, τη φτώχεια, τη δημογραφική κατάσταση που τροφοδοτούν όλη αυτή την κίνηση και αναμφισβητήτως αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου πολλά πράγματα έχουν γίνει για να οδηγήσουν σε μια σταθεροποίηση που φάνηκε να είναι πραγματική και από την άλλη μεριά βλέπει κανείς και το πόσο τεράστιο είναι το υπόβαθρο. Αυτέ είναι κάποιες σκέψει τώρα για την κατάσταση. Η διεθνής κοινότητα κάνει πολλά πράγματα, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη κάνει πολλές προσπάθειες και υπάρχουν βεβαίω ακόμα ορισμένα σημαντικά διακυβεύματα μέσα στην κατάσταση αυτή. Η κατάσταση στην Σαχέλ εδώ και πολύ καιρό λαμβάνει βοήθεια από τη διεθνή κοινότητα η οποία έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια. Πρόκειται για μια ζώνη όπου οι στατιστικές του Unique Aid λαμβάνει κατέτος 4 δισεκατομμύρια δολάρια που είναι σημαντικό ποσό ε, μεγάλο μέρος κατευθύνεται προς το Μαλί υπάρχουν επίσης και διμερείς βοήθειες επίσης πολλοί διεθνείς φορείς δραστηριοποιούνται η Ευρώπη με την ευρία έννοια το σύνολο των χωρών μελών και των θεσμικών οργάνων της Ενώσεως συμβάλλουν σε 40 περίπου τις 100 της βοήθειας αυτής. Από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως γνωρίζετε, υπήρξε σημαντική κινητοποίηση για την αντιμετώπιση της ε, κρίσης στο Μαλί. Το ίδιο και πιο πριν με μια στρατηγική για την Σαχέλ, με την έννοια να ληφθούν υπόψη οι περίπλοκες παράμετροι της ε, κατάστασης αυτής και η συμπληρωματικότητά τους με την ανάπτυξη που είναι ανέκαθεν σημαντικό επιδιωκόμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η διασύνδεση των δύο αυτών είναι και σίγουρα μία από τις παραμέτρους της κρίσης. Τώρα, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κινητοποιηθεί πολύ και σε μία διαδικασία που αποκλήθηκε η διάσκεψη των Βρυξελών για το Μαλί κινητοποίησαμε περίπου 2 δισεκατομμύρια ευρώ πριν από 2-2,5 χρόνια περίπου, έγιναν και επιχειρήσεις PSDC και στον Νίγηρα και στο Μαλή και για την εκπαίδευση στρατιωτικών με την ονομασία EUCAP Μαλί με κινητοποίηση πολλών χωρών μελών και με ένα αυξανόμενο ενδιαφέρον ομολογώ πολλών χωρών και ιδίως χωρών που είναι λιγότερο συνηθισμένα να έχουν σχέσεις με την υποσαχάρη Αφρική και που μπόρεσαν μέσα από επιχειρήσεις όπως η UTM να αναπτύξουν κέντρα ενδιαφέροντος σημαντικά. Εγώ μεταβαίνω συχνά σε χώρες μέλη όπου προσκαλούμε και που δεν είναι οι συνήθεις εταίροι και που θέλουν εκδηλώνουν ενδιαφέρον να κατανοήσουν καλύτερα και να συμβάλλουν καλύτερα στην αντιμετώπιση των διακυβευμάτων. Σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση εργάζεται επί της κινητοποίησης άλλων κονδυλίων στα πλαίσια διαφόρων περιφερειακών προγραμμάτων ύψους περίπου 3,5 δισεκατομμυρίων ευρώ για τα επόμενα χρόνια και σήμερα πάντως η Ευρωπαϊκή Ένωση συμπληρώνει την στρατηγική της με ένα σχέδιο δράσεως, περιφερειακής δράσεως που έχει το σημαντικό χαρακτηριστικό να εντοπίζει τέσσερις προτεραιότητες και εκεί να συγκεντρώνει τις δράσεις νέους, μετανάστευση, ε, ε, μεθοριακές ζώνες και ριζοσπαστικοποίηση. Αυτοί οι τέσσερις άξονες έχουν εντοπιστεί ως σημαντικά θέματα και επί των οποίων η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να προσφέρει μια σημαντική προστιθέμενη αξία λόγω και της ειδική γνώσης της. Τελειώνω λέγοντας ότι υπάρχει ένας αριθμός προκλήσεων που είναι οι πιο σημαντικές. Θα έλεγα πρώτα μιας περιφερειακής διάρθρωσης αντιμετωπίζουμε μια περιφερειακή κρίση με φορείς που είναι πάρα πολύ κατακαιρματισμένοι. Και εδώ παίζει ένα σημαντικό ρόλο η Αλγερία που είναι η μεγάλη δύναμη της περιοχής. Έχει δείξει και μέσω της στήριξης που έχει προσφέρει στην ε, διαδικασία συνομιλιών για το Μαλί ότι επιθυμεί να παίξει ένα σημαντικό ρόλο, σήμερα η Αλγερία έχει συνειδητοποιήσει πλήρως τη νέα περιφερειακή κατάσταση εδώ και αρκετά χρόνια και επιθυμεί να παραμείνει και στην εφαρμογή της διαδικασίας της Συμφωνίας του Αλγερίου ένας κέριος παράγοντας που μπορεί να συμβάλλει σε αυτήν την διάρθρωση όπου βέβαια παίζουν ρόλο και άλλοι ε, φορείς. Υπάρχει και μια πρόκληση αποτελεσματικότητας, αποδοτικότητας της διεθνούς βοηθείας. Πρόκειται για μια ζώνη η οποία ήδη δέχεται υψηλά ποσά βοήθειας. Το θέμα είναι να οργανωθεί καλύτερα, να εντοπιστούν καλύτερα οι προτεραιότητες, να δράσουμε πιο κοντά στις πραγματικότητες. Ο πρώτος ειδικός απεσταλμένος των ΗΕ για το Σαχέλ, ο κ. Ρωμάνο Πρόντι, ο οποίος υπέβαλε έκθεση προ 1,5 έτους περίπου, είπε ότι πρέπει να μπορέσουμε να δουλέψουμε διαφορετικά στη ζώνη αυτή. Είχε προτείνει τη δημιουργία ειδικού ταμείου Σαχέλ, όχι τόσο για να κινητοποιήσει κονδύλια, αλλά πιο διαθρωμένα. Πρότεινε επίσης να δημιουργηθούν προγράμματα έρευνας για την ζώνη Σαχέλ, είναι αλήθεια ότι υπάρχουν πολλές προκλήσεις και δεν είμαι βέβαιο ότι τις γνωρίζουμε τόσο καλά και τις προκλήσεις και τις πραγματικότητες. Τρίτο, βεβαίω κατά τη γνώμη μου υπάρχει και μια σημαντική πρόκληση σε ό,τι αφορά την οικονομική ανάπτυξη που να επιτρέπει να αναπτυχθεί η δημιουργικότητα και η απασχόληση. Εκεί αυτό θα βοηθήσει στην αντιμετώπιση και των προκλήσεων της μετανάστευσης, των νέων, Πρόκειται για ένα πληθυσμό νεότατο. Κάθε χρόνο εκατομμύρια νέοι μπαίνουν στην αναζήτηση εργασίας, στην αγορά εργασίας, στην αναζήτηση εργασίας, δεν βρίσκουν την θέση τους και σιγά σιγά μπορούν να φτάσουν μέσα από μια απόγνωση στις χειρότερες ε, παρεκκλήσεις. Κάτι το οποίο είναι και σύνηθες δυστυχώς για την νεολαία πολλών από τις χώρες αυτές και εκεί βεβαίως πρέπει να εγκύψουμε. Τέταρτο, πρέπει να επιτύχουμε τη σταθεροποίηση του Μαλή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει παρακολουθήσει και συνοδεύσει την υπογραφή της Συμφωνίας του Αλγερίου. Είναι βεβαίω περίπλοκη η κατάσταση. Παίζει το ρόλο του και ο Οργανισμός Ενωμένων Εθνών και η δύναμη Μίνους Μαλ. Πρέπει να ανταποκριθούμε και στις σημαντικές προσδοκίες που δημιουργεί η συμφωνία αυτή. Υπάρχει μεγάλη εμπιστοσύνη απέναντι στους Ευρωπαίους και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θεωρούμεθα ως από τους πιο θετικούς φορείς, επειδή γνωρίζουμε την ε, περιοχή, τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και οι χώρες μέλη από τις οποίες πολλές δραστηριοποιούνται στη ζώνη αυτή χαίρουν καλής ε, εκτίμησης, θετική εκτίμησης από τους ανθρώπους εκεί και αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να εγκύψουμε σιγά σιγά περισσότερο. Η πέμπτη πρόκληση είναι η απόσταση. Η διεθνής κοινότητα κινητοποιείται όταν υπάρχουν επίγουσες, έκτακτες καταστάσεις. Οι κίνδυνοι που προέρχονται από την Σαχέλ, χωρίς να θέλω να φαίνομαι απεσιόδοξος, είναι ακόμη μπροστά μας, δεν τις έχουμε αφήσει πίσω μας. Έχουμε 70-80 εκατομμύρια ανθρώπους που κατοικούν εκεί, σύντομα θα είναι 100 εκατομμύρια, αυτό είναι αναπόφευκτο, άρα πρέπει να γνωρίζουμε πώς θα οργανωθούμε για να αντιμετωπίσουμε το σύνολο αυτό των προκλήσεων υπό τις καλύτερες δυνατές συνθήκες. Και βέβαια να είμαστε και ως το δυνατόν πλησιέστερα στους Αφρου, Αφρικανούς παίκτες και φορείς που είναι επιτόπου. Γιατί υπάρχει κίνδυνος να μεγαλώσει η απόσταση ανάμεσα στην Ευρώπη και στην Αφρική γιατί η αντιμετώπιση δεν είναι πάντα ίδια για, απέναντι σε ένα κάπως παραδοσιακό Ισλάμ το οποίο αντιμετωπίζεται με κάποια δυσπιστία καμιά φορά. Δεν θα πρέπει να προκύψει μια έλλειψη κατανόησης μεταξύ των δύο πλευρών Ευρώπης και Αφρικής, ιδίως για την ε, ζώνη Σαχέλ. Τέλος, οι πολιτικοί, άνδρες και γυναίκες, οι κοινοβουλευτικοί μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο σε αυτές τις γέφυρες ανάμεσα στην Σαχέλ, την Αφρική και την Ευρώπη. Χρειαζόμαστε την συμβολή των πολιτικά υπεύθυνων, αυτοί να υποστηρίξουν όσο γίνεται περισσότερο οι διοικήσει. Ασφαλώ να τι κρίνουν εφόσον αυτό είναι αναγκαίο, αλλά χρειαζόμαστε και κάτι παραπάνω από αυτό κυκλοφορώντας σε διάφορες χώρες έχω την ευκαιρία να συναντώ εθνικούς βουλευτές που συχνά είναι πολύ ανοιχτοί και δείχνουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και επιθυμούν να πάνε όσο γίνεται πιο πέρα σε αυτό το ντοσιέ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε και εμείς πάρα πολύ. Κύριε Ρεβεράντε Ματών, διάφοροι συνάδελφοι έχουν ζητήσει το λόγο. Κύριε Αλιομαρή πρώτη. Παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Ντεμαντό για την διάγνωση που μας παρουσίασε. Βρήκα ότι ήταν πολύ ενδιαφέρουσα. Ακούγοντάς τον, είχα την εντύπωση πραγματικά πως το Σαχέλ έγινε και παραμένει μια γκρίζα ζώνη, όπως λένε και στρατιωτικοί, που δεν ε, κυβερνιέται μια επικίνδυνη περιοχή. Θέλω λοιπόν να σας κάνω δύο ερωτήσεις για να διευκρινίσουμε ακριβώς κάποια στοιχεία στο οποία αναφερθήκατε. Πρώτα απ' όλα, πέρα από τα χρήματα τα οποία πηγαίνουν ή θα πάνε στην περιοχή, τι άλλο κάνει συγκεκριμένα η Ευρωπαϊκή Ένωση για να ε, βοηθήσει στη διακυβέρνηση, για να μάθει τους ανθρώπους εκεί τη διακυβέρνηση και για να αντιμετωπίσει τα διάφορα λαθρεμπόρια όπλων, ναρκωτικών, ανθρώπων που έχουν άμεση σχέση με την τρομοκρατία. συνδέονται αυτά. Ιδιαίτερα για τα 3,5 δισεκατομμύρια που είπατε για τα επόμενα χρόνια, δώσατε κάποιο προσανατολισμό για το πού θα πάνε, αλλά θα ήθελα να γνωρίζω πιο συγκεκριμένα αν λαμβάνετε υπόψη αυτή η προβληματική που σας ανέφερα ή όχι. Έπειτα, σε πόσα χρόνια θα δαπανηθούν αυτά τα 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Δεύτερη ερώτηση. Αναφερθήκατε και είπατε πολλά για τη δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εγώ όμως θέλω να ξέρω συγκεκριμένα, με ακρίβεια, ποιες είναι οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίες βοηθούν και στις δράσεις άμυνας Μαλή, αν δεν απατώμε. Εμπλέχτηκαν πολλές χώρες εκεί και πόσες χώρες βοηθούν για τη σταθερότητα στην περιοχή. Ποιες άλλες χώρες παρεμβαίνουν. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Κύριε Γκόμες τώρα. Ευχαριστώ πολύ. Καλώς ήρθατε. Είπατε και συμφωνώ ότι η Αλγερία είναι μεγάλη δύναμη στην περιοχή, αλλά σε τι βαθμό το γεγονό ότι η Αλγερία και το Μαρόκο δεν μιλούν μεταξύ του, δεν συνεργάζονται εξαιτία ακριβώ τη δυτική Σαχάρα. αυτό δεν είναι ένα πρόβλημα στην όποια δράση, το ότι δύο αυτέ χώρε ενώ θα μπορούσαν να παίξουν σημαντικό ρόλο δεν το κάνουν. πέρα από το ότι γίνεται εκμετάλλευση της διαμάχης για τη Δυτική Σαχάρα, εσείς τι έχετε να πείτε για την νεότητα της Δυτικής Σαχάρας που ανυπομονεί. Θέλω να μου πείτε αν βλέπετε κάποια σχέση με όλες τις άλλες δυνάμεις που δρούν στην περιοχή, τρομοκρατία κλπ. Κάτι άλλο τώρα ανάμεσα σε εσά και την αποστολή σα και τον κύριο Μπεναντίνο Λεόν, ποια είναι η σχέση που είναι ο εκπρόσωπο του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για τη Λιβύη. Βλέπετε με τον ίδιο τρόπο κι εσείς και εμείς την κατάσταση στη Λιβύη ότι περιπλέκεται. Στο βορρά, ξέρουμε, οι περισσότεροι έρχονται από πιο κάτω από το Σαχέλ. Νιγηρία και λοιπά και φτάνουν στη Βόρεια Λιβύη και συνεχίζουν. Βλέπετε λοιπόν ότι η κατάσταση στη Λιβύη συνδέεται και με το πιο νότιο τμήμα και περιπλέκει την κατάσταση ακόμα περισσότερο πέρα από τα όπλα του Καντάφη που ξέρουμε που χρησιμοποιήθηκαν και οδήγησαν στη βία στο Μαλί κλπ. Τέλος, θέλω κι εγώ να ξέρω τι ακριβώς κάνουμε για την οικονομική ανάπτυξη, που είναι πολύ βασική για τη σταθερότητα στην περιοχή. Και για να συγκρατήσουμε τη μετανάστευση. Τι κάνουμε λοιπόν. Ευχαριστούμε ο κύριος Τσάρλς Τάνοκ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Συγχαρητήρια για τον ορισμό σας και από μένα σε μια περιοχή ιδιαίτερα επικίνδυνη και με πολλές προκλήσεις. Είχα την τιμή να συντάξω εδώ σχετική έκθεση στο Παϊκό Κοινοβούλιο, στην προηγούμενη θητεία δηλαδή για το Σαχέλ. Και πρέπει να σας ομολογήσω ότι είχα μπερδευτεί αρκετά, γιατί έπρεπε να ασχοληθώ και με το θέμα της Δυτικής Σαχάρας, που τελικά αποτέλεσε το κέντρο της έκθεσής μου, αντί να έχει το ίδιο βάρος με τα επικίνδυνα ζητήματα της τρομοκρατίας και το γενικότερο της σταθερότητας και της ευημερίας και της ασφάλειας στην περιοχή Σαχέλ. Τα θυμάμαι λοιπόν όλα αυτά και τις τελευταίες μέρες ξέρω ότι στο Τσάντ υπήρξε επίθεση το Βόρειο Μαλί εξακολουθεί να είναι κέντρο τζιχαντιστών. Διαβάζουμε επίσης τον τύπο ο Μπόκτα Ντελμόκτα, ο οποίος ηγήθηκε της ομάδας των Μουτζά. Υπήρξε μια συγχώνευση εκεί τρομοκρατικών ομάδων και φαίνεται ότι έχασε τη ζωή του από αεροπορική επίθεση που έγινε από τη Λιβύη. Βλέπουμε λοιπόν ότι όλες αυτές οι ομάδες είναι ιδιαίτερα ευκίνητες. Ο Μπέλματα ήταν και ο υπεύθυνο για τις τρομοκρατικές επίθεσεις ε, στην Αλγερία και φαίνεται ότι σκοτώθηκε από τις Αμερικανικές αεροπορικέ, δυνάμει. δεν είναι ακόμα σίγουρο, δεν έχει επιβεβαιωθεί. Οι διασυνδέσει συνεχίζονται και με τον Μπόκο Χαράμ στην Ιγυρία και νότια. Πάρα πολύ επικίνδυνο όλα αυτά. Και ακούμε ότι το λεγόμενο Ισλαμικό κράτος έχει παρουσία στην Λιβύη για να στηρίξει και άλλους σε άλλες περιοχές της Λιβύης που προσπαθούν να επιβάλλουν τη Σαριά. Εσείς λοιπόν πιστεύετε ότι στη ζωή σας ή τέλος πάντων στα 10 χρόνια πιστεύετε ότι θα μπορέσει και πάλι να λάβει χώρα το εκεί η κυρία Λοχμπίλερ. Ευχαριστώ, ευχαριστώ ιδιαίτερα κύριε Ρεβεράντε Μαντών. Έχω μία ερώτηση. Μιλήσατε για λαθρεμπόριο όπλων και ναρκωτικών. Θέλω να μιλήσουμε για το σώματεμπόριο. αν εξετάσετε την περιφέρεια Σαχέλ και το τι κάνει και η Ευρωπαϊκή Ένωση με τις ε, εξωτερικές σχέσεις, η ερώτηση που με ενδιαφέρει είναι τι ιδέες έχετε, τι μπορεί να κάνει κανείς εκεί διαφορετικά ή πώς μπορούμε να εντείνουμε τις προσπάθειές μας για να αντιμετωπίσουμε τη μάστιγα αυτή. Ευχαριστώ Πρόεδρε. και ο Σκάρβερ. Με την τραγωδία στις ακτές της Λιβύης και τον τραγικό αριθμό μεταναστών που πεθαίνουν Γιατί επικεντρώνεται το ενδιαφέρον στη Μεσόγειο για τους ανθρώπους, ενώ πολλοί πεθαίνουν και στη Σαχάρα, περνώντας Σαχάρα. Μήπως πρέπει να δούμε τι γίνεται και με αυτούς που πεθαίνουν προσπαθώντας να διασχίσουν τη Σαχάρα. Αυτούς λοιπόν που προσπαθούν να ισχύσουν τη Σαχάρα, θα του εξετάσουμε. Πριν φτάσουν στη Λιβύη, που πεθαίνουν προσπαθώντα να φτάσουν στη Λιβύη. Και πώ μπορούμε να του εμποδίσουμε και να του αποθαρρύνουμε να κάνουν αυτό το εξοδοτικό ταξίδι. Ευχαριστώ. Ο κύριο Πώς. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αναφέρατε, κύριε Πρέσβη, προκλήσει που αντιμετωπίζουμε στο Σαχέλ. Εννέα. Θα αναφέρω την Πέμπτη. Η αλλαγή του κλίματος είναι περίπλοκη και διασυνδέεται και με άλλα προβλήματα διαβίωσης, επιστημική ασφάλειας, μετανάστευσης και σύγκρουσης. Αντίθετα από το προσδοκόμενα, η βροχόπτωση από τη δεκαετία του 80 επαναλαμβάνεται, διαδέχεται την ξηρασία. Η βροχόπτωση δεν θα πρέπει να μας κάνει να εφησυχάσουμε, διότι έχουμε ακραία καιρικά φαινόμενα στο Σαχέλ και επηρεάζεται και η βλάστηση επιστημονικές αξιολογήσεις για την αλλαγή του κλίματος. Πώς πλήττει την περιοχή. Βρίσκω τα πορίσματα ότι δεν μου διαλύουν τα ερωτηματικά. Τι γίνεται με τους περιβαλλοντικούς πρόσφυγες που προσπαθούν να ξεφύγουν από τις δυσχερείς συνθήκες που δημιουργούνται λόγω της αλλαγής του κλίματος. Ευχαριστώ κύριο Σπαχνιού Κύριε Πρόεδρε, κύριε ειδική Εκπρόσωπε, αναφερθήκατε ακροθυγός στο θέμα της Μπόκο Χαράμ. Θα ήθελα να επανέλθω. Είναι πηγή ανησυχιών που όλο και αυξάνεται στην Νιγηρία αλλά και εκτός Νιγηρίας. Αφορά επίσης νομίζω και την Κεντρική Αφρική. Σύμφωνα με τις Νιγηριανές αρχές η Μπόκο Χαράμ έχει περίπου χίλιους μαχητές και οι ηγέτες της Μποκοχαράμ δήλωσαν πίστη προς την Τάις. και η επίθεση που έχει εκδηλωθεί εδώ και αρκετούς μήνες κατά διαφόρων γειτονικών χωρών όπως η Τσάντ, το Τσάντ υπάρχει στατιωτική αντιπαράθεση μεταξύ Μποκοχαράμ και στρατιωτικών δυνάμεων και δεν υπάρχει νίκη εναντί της Μπόκο Χαράμ όμως, παρά τις στρατιωτικές προσπάθειες. Και όλο και περισσότεροι μαχητές στηρίζονται από τη χρηματοδότηση της ΝΤΑΕΣ, μαχητές της Μπόκο Χαράμ. Πρέπει να εξετάσουμε αυτή την ε, χρηματοδότηση του ΝΤΑΕΣ στο Ιράκ. Αυξάνεται η χρηματοδότηση και υπάρχει και κάποια συνενοχή από πλευρά Ιρακινών αρχών σήμερα. Μπορείτε να μου πείτε περισσότερα. Αν υπάρχει συνενοχή από πλευράς Ιρακινού κράτους ε, όσον αφορά την ΤΑΕΣ και τη χρηματοδότηση. Τι σχέση μπορεί να έχει το ΤΑΕΣ με τους μαχητές της Μπόκο Χαράμ στην Νιγηρία. Ευχαριστώ. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Δεν θα ε, μπορούσα να απαντήσω εξίσου καλά σε όλες τις ερωτήσεις σας. Πρώτα απ' όλα γιατί ορισμένες ξεπερνούν την εντολή μου, αλλά και ορισμένες, όπως η τελευταία για παράδειγμα, με οδηγούν να πω το εξή, ότι στην εντολή μου δεν είναι τον Μπόκο Χαράμ αυτό καθεαυτό. Ε, βέβαια ασχολούμαι με την προβληματική αυτή, σε συναντήσεις όπου συμμετέχω, νομίζω ότι ο επόμενος επισκέπτης σας είναι πιο κατάλληλος για να σας απαντήσει σε αυτά. Βέβαια, η κατάσταση χαρακτηρίζεται από το παράλογο, από τον τρόπο με τον οποίο διαχέεται η Μπόκο Χαράμ. Ελπίζουμε Έχουμε τις ελπίδες μας δηλαδή στον νέο πρόεδρο της Νιγηρίας για να βάλει κάποια τάξη και να δούμε και πώς θα προχωρήσει η πολυμερής δύναμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία θα στηρίξει εκεί την κατάσταση. Πάντως, οι τρομοκρατικές ε, ομάδες που δρούν στην περιοχή είναι πιο παράλογες, λιγότερο οργανωμένες από ό,τι νομίζουμε, αυτή είναι και η δυναμία τους, αλλά είναι και μια δυσκολία για μας, γιατί είναι πιο δύσκολο να τις εντοπίσουμε και να έχουμε αποτελέσματα. Θα προσπαθήσω λοιπόν να απαντήσω τώρα και στην ερώτησή σας για την κλιματική διάσταση. Δυστυχώς οι ίδιοι Αφρικανοί ηγέτες δεν είναι αρκετά ευαισθητοποιημένοι. Ελάχιστα. Και είναι δύσκολο μαζί τους να προβλέψουμε μέτρα ή δράσεις για να αντιμετωπίσουμε τις κλιματικές αλλαγές. Υπήρξε το μεγάλο πράσινο τείχος, το οποίο αναφέρθηκε ο πρόεδρος της Ενεγάλης πριν από λίγο καιρό. Σε κάποιους θύλακες κάτι έγινε, αλλά δεν είχαμε δυστυχώς συστηματική πολιτική. Για τις αφρικανικές χώρες και τους αφρικανούς παράγοντες ε, είναι ένα θέμα μεταξύ πολλών άλλων, αλλά είναι πολύ δύσκολο να τους ευαισθητοποιήσουμε θύλακες υπάρχουν, υπάρχουν και κάποιες τραγικές καταστάσεις που δυστυχώς προστίθενται η μία στην άλλη και προσπαθούμε εντελώς κατακαιρματισμένα να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση στην περίπτωση του Τσάντ, με όλη την εξέλιξη στη λίμνη του Τσάντ προσπαθούμε να κάνουμε κάτι. Οι επιστήμονες πάντως να ξέρετε ότι και εκείνοι μεταξύ τους διαφωνούν πολλές φορές. Είμαστε στην αρχή της διαδικασίας. Επιθυμία μου είναι το τέλος της χρονιάς, το COP21, οι αφρικανικές χώρες, οι χώρες του Σαχέλ να βρουν τη θέση τους, να μπορέσουν να μιλήσουν και μπορούμε να φανταστούμε κάλλιστα να υπάρξει μια ειδική συνάντηση, ένα φόρουμ Σαχέλ. Προς το παρόν δεν προβλέπεται, αλλά για μένα θα ήταν μια καλή ιδέα να προχωρήσουμε με αυτόν τον τρόπο και έτσι να τους ε, αναγκάσουμε να συνειδητοποιήσουν πώς έχει η κατάσταση. Για το Σαχέλ πολλά είναι τα ερωτηματικά που συνδέονται πολύ περισσότερο με τη Σαχάρα αυτή καθ' αυτή παρά με το Σαχέλ. Και εξού και επανερχόμαστε στο ότι οι χώρες που βρίσκονται στο βορρά και στο νότο του Σαχέλ πρέπει να συνεργάζονται μεταξύ τους για να αντιμετωπίσουν μεταξύ άλλων και την πρόκληση αυτή την περιβαλλοντική που είναι κοινή για αυτούς. Υπήρξε μια οργάνωση πριν από μερικά χρόνια που ήταν το παρατηρητήριο για τη Σαχάρα και το Σαχέλ με έδρα την Τινησία. Επιστήμονες ανέλαβαν να, να δουλέψουν πάνω στα θέματα του ύδατος, των καλλιεργών, της προσαρμογής των καλλιεργιών, προσαρμογή του φυσικού πλούτου και αυτό που θέλουν είναι να στηριχθούν περισσότερο και να έχουν περισσότερους συνομιλητές. Πολλές ερωτήσεις σας έχουν να κάνουν με το λαθρεμπόριο, με το εμπόριο ανθρώπων, τη μετανάστευση. Όντως, την πραγματικότητα αυτή της Σαχάρας, δηλαδή των ανθρώπων που διασχίζουν τη Σαχάρα για να μεταναστεύσουν, δεν είναι τόσο γνωστή. Σίγουρα υπάρχουν πολύ περισσότερα δράματα και δυσκολίες από ό,τι γνωρίζουμε μέχρι τώρα. Ο κύριος προσανατολισμός έχει να κάνει με περισσότερη συνεργασία μεταξύ των χωρών της περιοχής, ώστε να συνεργαστούν μαζί μας και να λάβουν υπόψη τους την πραγματικότητα. Μία από τις δυσκολίες που έχουμε είναι ότι ε, το Σαχέλι αποτελεί ένα κρίκο, ένα μικρό κρίκο μάλιστα της όλης αλυσίδας. Η διαδικασία του Ραμπάτ όπου συμμετέχουν χώρες της Βόρειας Αφρικής, ε, της Δυτικής ε, και του Κέντρου, ίσως είναι μια σωστή κλίμακα. Αν έχουμε μια πιο μεγάλη, είναι δύσκολο να βρούμε συγκεκριμένες δράσεις για να βοηθήσουμε. Σήμερα λοιπόν θέλουμε να δουλέψουμε για τον έλεγχο, την πρόληψη. Εδώ και πολύ καιρό γίνεται έλεγχος στα αεροδρόμια, ενισχύεται δηλαδή από τον ένα χρόνο στον άλλο. Υπάρχει συστηματική συνεργασία στον τομέα αυτό σήμερα. Πολύ γρήγορα όμως ερχόμαστε αντιμέτωποι με το πρόβλημα της ανεργίας των νέων. Γίνονται εκστρατείες ενημέρωσης. Κάποια αποτελέσματα δίνουν. Δείχνουμε ποια είναι η δυσκολία δηλαδή της μετανάστευσης, ποια είναι η δυσκολία να βρει κανείς δουλειά στις χώρες του Βορρά. Βέβαια δεν είναι τόσο αποτρεπτικά όλα αυτά όσο θα θέλαμε, Κάποιοι έλεγχοι επιτόπου έχουν δώσει αποτελέσματα μέχρι τώρα. Με τις πυρόγες που φεύγαν από τη Μαυριτανία ή τη Σενεγάλη προς τα Κανάρια νησιά. Καταφέραμε να ελέγξουμε αρκετά αποτελεσματικά αυτές τις περιπτώσεις. Αλλά βέβαια από την άλλη ξέρουμε ότι η δημογραφική κατάσταση είναι ιδιαίτερα περίπλοκη και έχει να κάνει με την κακή εξίσωση, κατάρτιση και θέσεις απασχόλησης η κοινωνική κατάσταση είναι τέτοια που η κοινωνία κινείται. Η μετανάστευση γίνεται και προς την Αφρικανική Ήπειρο, τις χώρες της Βόρειας Αφρικής. Βέβαια ούτε το 10% από τη Δυτική Αφρική δεν πηγαίνει στην Βόρεια Αφρική θέλει να προχωρήσει κι άλλο. Ε, αυτό δηλαδή που πρέπει να γίνει είναι να δουλέψουμε με τους νέους, να τους βοηθήσουμε να βρουν δουλειά επί τόπου. Ίσως αυτοί που θέλουν να επιστρέψουν να μπορούν να έχουν κάποια βοήθεια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πριν από χρόνια στήριξε ένα πρόγραμμα στο Μαλί, ένα κέντρο κατάρτισης δηλαδή και ενημέρωσης για την μετανάστευση. Ενημέρωνε δηλαδή τους κατοίκους του Μαλή. Αλλά αυτή είναι μια διαδικασία πολύ μακροχρόνια. Χρειάζεται συνεργασία με τις αφρικανικές χώρες και σε περιφερειακό επίπεδο αλλά και με κάθε χώρα χωριστά. Στην Αμπούσα πριν από λίγε μέρες και όσα ασχολείται γιατί είναι θέμα και ελεύθερη κυκλοφορίας στη Δυτική Αφρική του πληθυσμού εκεί. οι χώρες της Δυτικής Αφρικής, όχι οι χώρες Δυτικής Αφρικής θέλουν διάλογο μαζί μας. Για να συζητήσουμε για τη μετανάστευση στη Σαχέλ και πέρα τη Σαχέλ. Θέλω να πω ότι υπάρχει συνειδητοποίηση όλο και περισσότερο μεταξύ των χωρών της περιοχής και οι διάφοροι αξιωματούχοι αλλά και οι ηγέτες καταλαβαίνουν ποια είναι η πρόκληση, ποια είναι η κίνδυνη. Η δουλειά όμως είναι μακροπρόθεσμη. Πολλές χώρες προσπάθησαν να βρουν κάποια λύση με περισσότερη ή λιγότερη επιτυχία. Ο δρόμος είναι μακρύς. Ο έλεγχος στη Σαχάρα είναι αναγκαίος. Πρέπει να ενισχύσουμε τους χώρους από όπου φεύγουν οι μετανάστες, από όπου ξεκινούν πρώτα απ' όλα. Περιορισμένα μέτρα έχουν ληφθεί μέχρι τώρα που δεν έχουν εμποδίσει τη μετακίνηση. Μπορεί να την έχουν περιορίσει σε ένα βαθμό. Υπάρχουν και ειδικοί, ειδικά όργανα των Ηνωμένων Εθνών που βοηθούν, που βοηθούν και στον επαναπατρισμό όσων θέλουν να επιστρέψουν. Το θέμα το γιο, της γεωστρατηγικής του Σαχέλ και της Δυτικής Αφρικής είναι κεντρική σημασίας. Η λογική είναι να έχουμε μια μακρόχρονη οπτική η τρομοκρατία, το λαθρεμπόριο κτλ. γίνονται σε μεγάλη κλίμακα, δίχως άλλο. Αυτή τη μεγάλη κλίμακα πρέπει να αντιμετωπίσουμε με μια δράση σε εξίσου μεγάλη κλίμακα. Γιατί αν θέλουμε να δράσουμε και στη Βόρεια Αφρική και στη Δυτική Αφρική είναι πολύ δύσκολο. Πρέπει να προσπαθήσουμε να οριοθετήσουμε, να περιορίσουμε τη δράση μας σε διαδρομές, σε συγκεκριμένα φαινόμενα και αυτά να αντιμετωπίσουμε κατά περίπτωση. Να συμφιλιώσουμε δηλαδή μια προσέγγιση συνολική με την αναγκαιότητα να δράσουμε επιτόπου. Τώρα για τις σχέσεις Αλγερίας και Μαρόκο είναι στρατηγική σημασίας. Ιδεοδός, μια τέτοια συνεργασία θα βοηθούσε πολύ. Αλλά αντιλαμβανόμαστε ότι εντάσει που υπάρχουν ανάμεσα στις δύο χώρες εμποδίζουν μια τέτοια συνεργασία. Και καθένας πετάει το μπαλάκι στον άλλον, το ξέρουμε. Βόρειο Μαλή και Δυτική Σαχάρα. Θα έπρεπε να ασχοληθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είμαι εγώ αρμόδιος. Ορισμένοι πιστεύουν πω ναι. Ξέρουμε ότι υπάρχει διάσταση απόψεων. Μεγάλη. Ίσως ήρθε η στιγμή να πούμε Ας συγκεντρώσουμε τις προσπάθειές μας όλες οι ευρωπαϊκές χώρες με τα Ηνωμένα Έθνη. Έτσι μπορούμε να πιέσουμε μέχρι τέλους και έτσι να βοηθήσουμε να λυθεί το πρόβλημα. Κρατάει πάρα πολύ το πρόβλημα εκεί. Ίσως ήρθε η στιγμή να αλλάξουν τα πράγματα μια και έξω. Δυτική Σαχάρα και Βόρειο Μαλή έχουν σχέση και διασύνδεση το εντοπίσαμε πριν από λίγο καιρό. Δύσκολο βέβαια να πει κανείς ποια ακριβώ είναι. Οι Μαροκινοί πέταν τον μπαλάκι στο μαλλί και αντίστροφα. Είναι δύσκολο. Επαφές υπάρχουν, κοινωνιολογικά υπάρχουν διασυνδέσεις, ίσως όσο τόσο μεγάλες τώρα. Η Λιβύη, όπως και το Μποκοράμ δεν είναι στην δικιά μου εντολή, οπότε δεν έχω να σας δώσω πληροφορίες. Παρακολουθούμε τα γεγονότα και παρακολουθούμε και τις προσπάθειες που κάνει ο Μπερναντίνο Λεόν γι' αυτό. Το θέμα τώρα της οικονομικής ανάπτυξης είναι ζωτική σημασία, είναι προς το συμφέρον της διεθνούς κοινότητας. Εδώ και μερικά χρόνια είχαμε την, ε, μια προσέγγιση αντοχής, δηλαδή ε, θέλαμε να αποφύγουμε τον κίνδυνο βραχυπρόθεσμα και είπαμε ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί το ενδεχόμενο μια άμεσης καταστροφής, ανθρωπιστικής. Θελήσαμε να ενισχύσουμε μια τοπική γεωργία, μια τοπική κτηνοτροφία, τοπικά, για να μπορεί ο κόσμος στην καθημερινότητά του να έχει αυτά που του χρειάζονται. Αυτά βέβαια δεν φτάνουν για να υπάρξει μια γενικότερη οικονομική ανάπτυξη. Εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα θέμα το οποίο κατά την προσωπική μου γνώμη δεν αντιμετωπίζεται σωστά. Έχουμε ασχοληθεί τα τελευταία χρόνια με τις υποδομές, τις ενεργειακές, αλλά λιγότερο με τη γεωργία που θα μπορούσε να προσφέρει πολλές θέσεις απασχόληση. Πιστεύω επίσης ότι η δημιουργία επιχειρήσεων, το να αναπτυχθεί ο ιδιωτικό τομέα, επιχειρήσεις μικρές, μεγάλες, ε, επίσημε, λοιπόν, είναι το στοιχείο κλειδί. Η διεθνή κοινότητα θα έπρεπε να ασχοληθεί περισσότερο με αυτό. Να αναπτυχθεί δηλαδή ο ιδιωτικό τομέα. Να ψάξουμε να βρούμε επιχειρηματίες. Υπάρχουν στην Αφρική, μπορεί να μην είναι πολύ άριθμοι και κυρίω αντιμετωπίζουν ένα σωρό προβλήματα, διαφθορά, γραφειοκρατία. Θα έπρεπε να του στηρίξουμε περισσότερο. Οι ευρωπαϊκές χώρες ποιες δρούν. Τρεις είναι οι χώρες που συνεισφέρουν στη Μινουσμά. Οι κάτω χώρες, η Δανία και η Σουηδία. Πολλές ευρωπαϊκές χώρες συμμετέχουν στο UTM, e είναι οι περισσότερες. Και οι χώρες που δεν δραστηριοποιούνταν πολύ, Πολωνία για παράδειγμα, Τσεχία, Ρουμανία, μιλάω για αυτές γιατί είχα άμεσα επαφές, ήρθαν και με βρήκαν, μου ζήτησαν να συζητήσω μαζί τους και οι βαλτικές χώρες. Οι χώρες αυτές λοιπόν ανακάλυψαν τι διακυδεύεται σε αυτό το τμήμα του κόσμου και θέλουν να δραστηριοποιούνται στην περιοχή. Αλλιώς υπάρχουν κανένα δεκαριά ευρωπαϊκές χώρες οι οποίες παραδοσιακά δρουν. Η Ισπανία παίζει σημαντικό ρόλο, η Πορτογαλία, Βέλγιο, Λουξεμβούργο. Έχουμε δηλαδή έναν δυνατό πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θέλει να δραστηριοποιείται όλο και περισσότερο, που στηρίζει τη δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και είναι ένας κύκλος που μεγαλώνει σε μια περιοχή που ορισμένοι μόλις τώρα ανακαλύπτουν. Η δράση για τη διακυβέρνηση τώρα. Αυτή είναι μια από τις μεγάλες δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περιοχή καλύπτει πολλά πράγματα. Ο κύριος άξονας τα τελευταία δέκα χρόνια ήταν η αποκέντρωση. Μεταρρύθμιση σε τοπικό επίπεδο, πιο κοντά στον κόσμο. Συνεργασία για την αποκέντρωση με τη Γαλλία για παράδειγμα, κάτι το οποίο άλλαξε αρκετά την κατάσταση γιατί οι τοπικές αρχές, οι δίκες ήρθαν πιο κοντά στον κόσμο. Υπάρχουν μεταρρυθμίσεις και στη δικαιοσύνη, πιο δύσκολες, ευάλωτες ακόμα. Δυσκολεύονται ακόμα οι χώρες αυτές με τη διαφθορά. Είναι μια σημαντική μάστιγα που παίζει ρόλο, απογοητεύει τον κόσμο. Τον κάνει να χάνει το ηθικό του. Κατά τα άλλα η δίκηση στηρίζεται κατά περίπτωση του Υπουργείο Άμυνας, Εσωτερικών. Συνολικά έγιναν πολλά πράγματα. Αυτό που είναι αλήθεια είναι ότι πολλές αφρικανικές χώρες δεν κατάφεραν να βρουν την ισορροπία τους στις σχέσεις με τον κόσμο. Δεν θα έλεγα ότι όλοι νιώθουν όπως θα έπρεπε να νιώθουν μέσα σε μια χώρα. Είναι το θέμα της ηθαγένειας, των δικαιωμάτων του πολίτη. Εκεί υπάρχει αδυναμία. Παρά τα όσα έγιναν. Που, την εκπαίδευση που μαθαίνουμε στα παιδιά, ποια είναι η χώρα τους, τι είναι η χώρα τους. Γίνεται δουλειά. Στον τομέα της συγκέντρωσης. 52% έχουμε δράσει Ευρωπαϊκής Ένωσης εθνικά προγράμματα που έχουν να κάνουν με τη διακυβέρνηση. Όντω πολύ γρήγορα βέβαια φτάνουμε σε ευαίσθητα πολιτικά ζητήματα κάθε φορά. Και ακριβώ εδώ είναι που δεν ξέρουμε πώς να δράσουμε. Έχουμε και πολλές ε, δράσεις δημοσιονομικές. Αυξήθηκε ο προπολογισμό τα τελευταία χρόνια και βασιζόμαστε σε κριτήρια που έχουν να κάνουν με το κράτος δικαίου, κύρια, με το σεβασμό της χρηστής διακυβέρνησης, την τήρηση των κανόνων, της νομιμότητας, των μεταρρυθμίσεων σε βάθος, ακόμα και αν σήμερα το κράτος δικαίου μένει να είναι ένα σπαράγοντας και πολιτιστικός. Πρέπει δηλαδή να περάσει πρώτα μέσα από την οτροπία των ανθρώπων στις χώρες αυτές. Το λαθρεμπόριο είναι ένας από τους τομείς σχετικά με τους οποίους δεν κάνουμε πολλά ακόμα. Παραμένει αρμοδιότητα χωρών, των ίδιων των χωρών. Συνεργασία της αστυνομίας, ναι. Σήμερα έχουμε τη UCAP και έτσι σιγά σιγά καταρτίζοντας ομάδες της αστυνομίας κάνουμε περισσότερα. Δεν πρόκειται μόνο για το Σαχέλ. Οι αστυνομικοί είναι οι πρώτοι που λένε ότι αν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε το λαθρεμπόριο στο Σαχέλ, πρέπει να το αντιμετωπίσουμε πρώτα απ' όλα στην ε, Νέα Μπισάου ή στα λιμάνια, δηλαδή από εκεί που μας έρχονται. Το να αντιμετωπιστεί το λαθρεμπόριο στην έρημο, ε, σίγουρα δεν είναι ότι το πιο εύκολο. Πάντως υπάρχει η βούληση σήμερα να προχωρήσουμε. Τα 3,5 δισεκατομμύρια προβλέπονται για μέχρι το 2020. Ελπίζω να απάντησα στις πολυάριθμες ερωτήσεις σας, οι οποίες ήταν όλες πολύ συγκεκριμένες και σωστές. Ευχαριστώ πολύ κύριε Ντεμεντών. Ευχαριστώ πολύ για αυτή τη συνάντηση. Σας ευχόμαστε καλή τύχη. Σας ευχαριστώ.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 So, uh, colleagues, let's proceed. Ας προχωρήσουμε, συνάδελφοι. Θα γίνει ανταλλαγή απόψεων με κάποιον που έρχεται συχνά στην Επιτροπή μας και την Υποεπιτροπή μας ε, Άμυνας, ο κύριος Ζιλ Ντεκέρκοφ λοιπόν. Είναι ο συντονιστής αντιτρομοκρατικής δράσης Ευρωπαϊκής Ένωσης και θέμα της συζήτησης είναι η τρέχουσα κατάσταση όσον αφορά τη συνεργασία με τρίτες χώρες ένας τομέας σημαντικότατος, όπως γνωρίζετε, διότι χρειαζόμαστε τη συνεργασία τους αν θέλουμε να ελέγξουμε το φαινόμενο. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι ξανά εδώ. So that we can have uh, Για να είμαι σύντομος και να έχουμε ανταλλαγή απόψεων και ερωταπαντήσεις, θα ήθελα να παρουσιάσω το πώς εφαρμόζεται η δήλωση των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων μετά τις επιθέσεις στο Παρίσι που έλαβαν χώρα στις 12 Φεβρουαρίου εμπεριείχε ε, τρεις πτυχές ε, και θα επιμείνω επί της τρίτης πτυχής καταστολή. Οι ήπιες πολιτικές αποκαλώ, αλλά είναι φιλόδοξες, δεν είναι πολύ ήπιες και ε, εξωτερική διάσταση. Όσον αφορά το πρώτο καλάθι του ΣΥΠΗΝ, οι Υπουργοί Εσωτερικών και Δικαιοσύνης θα το συζητήσουν αύριο στο Λουξεμβούργο πώς έχουμε προχωρήσει όσον αφορά το διαδίκτυο, τέτοια θέματα, διαχείριση συνόρων, κυρίως να εντοπίσουμε ε, την διακίνηση υπόπτων για ότι είναι ξένοι μαχητές, ε, εμπόριο ε, όπλων, δικαστική ανταπόκριση. Θα ξεκινήσω αναφερόμενος τα τρία καλάθια που ανέφερα αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων. Πρέπει να κινηθούμε σε αυτού του τομεί. Για το διαδίκτυο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ξεκινήσει με το τέλο του έτου ένα φόρουμ, ένα βήμα συζητήσεων για να συζητηθούν όλε οι πτυχέ. Έλεγχο του διαδικτύου, επιτήρησή του, πώ μπορούμε να αφαιρέσουμε παράνομο περιεχόμενο από το διαδίκτυο. Η Ευρωπόλ από 1η Ιουλίου σχετικά με αυτό θα δημιουργήσει μια συγκεκριμένη μονάδα για το διαδίκτυο για να εντοπίζει όλο και περισσότερο παράνομο περιεχόμενο ε, και να το επισημαίνει σε εταιρείε του διαδικτύου και να αναπτύξουμε, αναπτύσσω εγώ αυτή την πτυχή και εξωτερικά τα αντίμετρα και κάτι που δεν ξεκίνησε αλλά πρέπει να εξεταστεί. Η κρυπτογράφηση που πρέπει να χρησιμοποιείται στις εταιρείε του διαδικτύου για να αντιμετωπιστούν φαινόμενα του τύπου του Snowden Leaks. Για τη διαχείριση των συνόρων η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ολοκλήρωσε μόλις τώρα κοινού δείκτες κινδύνου ούτω ώστε οι μεθοριοφύλακε στα εξωτερικά σύνορα τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω να ελέγχουν του πολίτε τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω όταν διασχίζουν τα εξωτερικά σύνορα με τον ίδιο τρόπο η νομοθεσία δεν επιτρέπει συστηματικό έλεγχο των πολιτών τη Ευρωπαϊκή Ενώσεων όταν διέρχονται τα εξωτερικά σύνορα, όταν απέρχονται και όταν επιστρέφουν. Αλλά θα πρέπει να έχουμε μεγαλύτερο συντονισμό. Καλύτερη συστηματική προσέγγιση. Προχωρούμε. Άλλη πτυχή, σημαντικότατα για να εντοπίσουμε ύποπτου ταξιδιώτε, που ανελημμένα το ανέφερα στο Ευρωκοινοβούλιο και γνωρίζει το θέμα του Ευρωκοινοβούλιο, τη σημασία που δίδει το Συμβούλιο όσον αφορά τους φακέλους, στα αρχεία PNR, των προσωπικών στοιχείων των επιβατών, ε, υπό αυστηρέ συνθήκε και ρήτες διαφύλαξη για την προστασία της ιδιωτικής ζωής θα πρέπει η κοινότητα επιβολή του νόμου να έχει πρόσβαση στο PNR, διότι όπως ανέφερα επανειλημμένα, οι υπηρεσίε ασφαλείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σε θέση να εντοπίζουν 70 με 80% των ενδεχομένων των πιθανών τζιχαντιστών στην καθημερινή τους δουλειά, αλλά έχουμε 20 με 30% των επιδόξων τζιχαντιστών που μπορούν να αναχωρήσουν χωρίς να το πιστούν. Το PNR είναι ένας τρόπος, από τους λίγους τρόπους, μη πω ο μοναδικός, για να εστιάζουμε καλύτερα τις προσπάθειές μας να εξετάζουμε λοιπόν τον τεράστιο αριθμό των επιβατών για να εντοπίσουμε του υπόπτου. Τρίτον, ε, επιμερισμό των πληροφοριών. Πώ οι αστυνομικέ αρχέ και οι υπηρεσίε ασφαλεία των κρατών μελών μπορούν να μοιράζονται περισσότερο τι πληροφορίε με το Eurojust και την Europol και τη Frontex. Πώ μπορούμε καλύτερα να δίνουμε πληροφορίε στο σύστημα πληροφοριών του Σέγγεν, να δίνουμε στοιχεία στι διάφορε διάβλους επικοινωνία τη ε, Interpol, προσπαθούμε και να αντιμετωπίσουμε το θέμα. Εμπόριο όπλων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο Ευρωπαϊκό Θεματολόγιο για την Ασφάλεια ανακοίνωσε ότι θα υποβάλει σχέδιο νομοθεσία για την εναρμόνιση, καλύτερη εναρμόνιση των μέτρων και να είναι πιο αυστηρά τα μέτρα και οι προδιαγραφές για τον αφοπλισμό ε, των ε, πυροβόλων όπλων και γίνεται προσπάθεια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για νομοθεσίε τη Ευρωπαϊκής Ένωσης για να εναρμονίσουμε την συμπεριφορά των ατόμων που αποχωρούν την Ευρωπαϊκή Ένωση για να εκπαιδευτούν για το τζιχάντ και για να επιστρέψουν. Ε, θα εφαρμόσουν συλλογικά τα 28 κράτη-μέλη μέσω εργαλείου της Ευρωπαϊκής Ένωση. Ε, ε, ε, αυτά που λέει το ψήφισμα το ΙΕ 2178 για το θέμα τζιχαντιστών και άλλο σημαντικό θέμα πως συλλέγουμε στοιχεία αποδείξεις ότι κάποιος πολεμούσε στις α, γραμμές του Ντάες ε, στην Τζαμάτα Ρούστρα ή κάπου αλλού εφόσον δεν συνεργαζόμαστε με το καθεστώς Αζάντ πώς τους εντοπίζουμε, πώς τα αποδεικνύουμε πρέπει να αφήνουν ηλεκτρονικά ίχνη αυτοί οι άνθρωποι ότι συμμετέχουν σε τρομοκρατική οργάνωση. Αν δεν έχουν τέτοια ίχνη δεν υπάρχουν αποδείξει για να δικαστούν. Χρειάζονται συγκεκριμένε ρυθμίσει και διευθετήσει, ρυθμίσει με του Αμερικανού φίλου. Διότι περισσότερε εταιρείε του διαδικτύου είναι Αμερικανικέ, Οπότε υπάρχουν πολλά αιτήματα που υποβάλλουν διάφοροι φορεί και οι δικαστέ στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να έχουν πρόσβαση σε διεύθυνση internet provider και να συλλέξουν ηλεκτρονικά στοιχεία. Αυτά είναι στο πρώτο καλάθι. Το δεύτερο καλάθι τώρα ε, αφορά την Επιτροπή σας. Είναι η ήπια απάντηση που περιέχεται εδώ. Αλλά πώς μπορούμε να εμποδίσουμε την τρομοκρατία εν πρώτης, τη ριζοσπαστικοποίηση, ε, πώς καταπολεμούμε αντισημιτικά και ισλαμοφοβικά θέμα, ομιλίες και συμπεριφορές. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, καταβάλει προσπάθειες, ότι πρόεδρος Τίμερμανς ε, πρόκειται να διοργανώσει την 1η και 2η Οκτωβρίου μεγάλη διάσκεψη όσον αφορά αυτά τα θέματα, τις προκλήσεις αυτές που αντιμετωπίζουμε, Ισλαμοφοβία και αντισημιτισμό. Ε, διερευνούμε με διάφορους επιτρόπους το πώς μπορούμε αυτές τις ανησυχίες να τις εντάξουμε όλο και περισσότερο σε διάφορα προγράμματα χρηματοδοτήσεις για την νεολαία, για την παιδεία, για τον αθλητισμό, για ε, τον πολιτισμό. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Έχουμε δημιουργεί ένα κέντρο αριστείας στο δίκτυο για τη ριζοσπαστικοποίηση. Όσο βλέπουμε, όσο ταξιδεύουμε συγχώς που αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα της νομοκρατίας, μας ζητούν να το στηρίξουμε στην, στον τομέα της προλήψεως. Και είναι σημαντικό εμείς οι ίδιοι να είμαστε καλά οργανωμένοι και να έχουμε τη δυνατότητα να στείλουμε εμπειρογνώμονες. Έχουμε το δίκτυο ευαισθητοποίησης για τη ριζοσπατικοποίηση και είναι ένα θέμα για... που πρέπει να γίνει πιο καλά διαθρωμένο και θα μας βοηθήσει κάτι τέτοιο. Ξεκινήσαμε συνεργασία με την Ιορδανία και με το Μαρόκο και με την Τινησία που ζητούν υποστήριξη να τους βοηθήσουμε να σχεδιάσουν στρατηγικές και να εφαρμόσουν μια στρατηγική προληπτική θέλουμε να βοηθήσουμε τις χώρες να κινηθούν καλύτερα στο μέλλον και κάτι άλλο σαν αφορά αυτή την ήπια ανταπόκριση που αφορά περισσότερο Μεσογείου πώς αντιμετωπίζουμε την επιστροφή εκείνων που πολέμησαν στη Συρία και το Ιράκ. Όπως είπα είναι πρόκληση καμιά φορά για να τους δικάσουμε δεν έχουμε τα στοιχεία και δεν μπορούμε να τους παρακολουθούμε καθημερινά 24 ώρες 24 ώρες είναι πολύ απαιτητικό όσον αφορά τους ανθρωπίνους πόρους. Και εγώ απευθύνω έκκληση στους Υπουργούς Δικαιοσύνης να δημιουργήσουν προγράμματα απεμπλοκής δεν ξέρω, επανένταξη θα τα αποκαλέσουμε από ριζοσπαστικοποίηση. Πρέπει να αναπτύξουμε περισσότερο αυτό που ξεκίνησα κάποια κάτι μέλη. Το Channel στο Ηνωμένο Βασίλειο, Exit στη Γερμανία, ένα πρόγραμμα στο Άρχους στη Δανία. Χρειαζόμαστε όμως κάτι πιο στέρεο και ε, η κυρία, ε, η Επίτροπος για τα θέματα δικαιοσύνης ασχοληθεί με αυτό το θέμα και το φθινόπωρο θα διεξαχθεί μια διάσκεψη για να συλλεχθούν οι βέτησες πρακτικές και να δούμε πώς θα κινηθούμε. Τρίτο καλάθι που αφορά μέσα την Επιτροπή σας, που είναι η εξωτερική πτυχή στο τρίτο αυτό καλάθι. Θα θυμόσαστε ότι στις 9 Φεβρουαρίου, και αυτό ήταν ένα από τα δομικά στοιχεία που οδήγησε στη δήλωση των αρχηγών Κατών κυβερνήσεων, το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων υιοθέτησε άκρος φιλόδοξα συμπεράσματα που σε μία φράση ε, οδηγούσαν σε μεγαλύτερη, πολύ μεγαλύτερη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ενώσεως στην άμεση γειτονία της. Από Μαρόκο μέχρι Τουρκία, τα Βαλκάνια, όσον αφορά την ασφάλεια και την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Βλέποντας τα συμπεράσματα πρέπει να ομολογήσω ότι είναι πολύ απαιτητικά για την εξωτερική υπηρεσία δράσης, για τους συναδέλφους μου και εμένα και ξεκινήσαμε την εφαρμογή των συμπερασμάτων. Θα διατρέξω τα διάφορα σημεία των συμπερασμάτων, τις ιδέες, 8-9 ιδέες. Α, θέλουμε να αναπτύξουμε πιο στοχευμένο διάλογο για την ασφάλεια και την καταπολέμηση τρομοκρατίας. Δεν θέλουμε μόνο διάλογο με τους ομολόγους μας εξωτερικών υποθέσεων των Υπουργείων Εξωτερικών των χωρών, θέλουμε να μιλήσουμε και με, το, με εκείνους που είναι επιφορτισμένοι με την κατανοήση τρομοκρατίας, υπηρεσίες ασφαλείας, επιβολής του νόμου, δικαστικ, βασικός κλάδος των χωρών. Ε, θα πρέπει όλες τις πλευρές ε, θα πρέπει όσοι πλευρές συμμετάσχουν, οι θεσμοί τη Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωπόλου, η η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Frontex, ε, υποφαινόμενο και οι συνάδελφοι της υπηρεσίας εξωτερικής Δράση. Δεν έγινε η πρώτη συνάντηση λόγω κάποιων διαφορών. Όχι τόσο επί της ουσίας, είχαμε διαφωνήσει με το Μαρόκο για άλλο θέμα και με την Τινησία ανεβλήθησαν οι συνομιλίες γιατί έγιναν επισκέψεις υψηλότερου επίπεδου, επισκέφθην με, με τον Προεδρεύοντα του Συμβουλίου την Τινησία, κυρία Μογκερίνη, συνάντησε επανειλημμένα τον Πρωθυπουργό, ο Πρωθυπουργός ήρθε στις Βρυξέλλες και Κάναμε κάποιε προτάσει στον Πρωθυπουργό τη Τινησία για να τον βοηθήσουμε να αντιμετωπίσει τι τεράστιε προκλήσει που αντιμετωπίζει η χώρα όσον αφορά την τρομοκρατία. Σύντομα θα γίνει συνάντηση με το Λίβανο, με την Τουρκία και ελπίζουμε και με το Μαρόκο ακόμα φέτο και την Τινησία και την Αλγερία για φέτο. Μετά, θέλουμε να διερευνήσουμε με όλε τις χώρες αυτές και τα Υπουργεία τους τα αρμόδια ποιες είναι οι πραγματικές τους ανάγκες. Ξεκινήσαμε με ένα εργαστήριο με... στο Λίβανο. Όλοι οι φορείς του Λιβάνου ήταν παρόντες. Ενδιαφέρουσα, πολύ ενδιαφέρουσα εμπειρία ήταν παρόντα τα κράτη-μέλη μέσω των αστυνομικών αρχών, των διοκτικών αρχών των χωρών εντοπίσαμε τι ο τρόπος ακριβώς πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τη χώρα να βρει απαντήσεις. Κυρίως θέλουμε να βοηθήσουμε τις χώρες να εφαρμόσουν ε, το ψήφισμα 2178 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΙΕ που προανέφερα. Ξεκινήσαμε από το Λίβανο. Θα είμαι στην Τουρκία την επόμενη εβδομάδα για την ίδια προσπάθεια. Ελπίζουμε ε, να γίνουν οι επαφές αυτές πριν το καλοκαίρι και μετά την Ισία, Μαρόκο, Αίγυπτος, Ιορδανία το 2015 και Αλγερία του χρόνου. Έτσι θα φτάσουμε στην τρίτη πτυχή, δηλαδή να αναπτύξουμε αντιτρομοκρατικά σχέδια δράσης. Θα πείτε γιατί κινείστε σε ξεχωριστές πορείες όταν συζητούμε με αυτές τις χώρες όσον αφορά τις εταιρικές συμφωνίες. Λόγω της σημασίας και της κατεπίγουσας ανάγκης να αντιμετωπιστεί η απειλή, θέλουμε να έχουμε συγκεκριμένο έγγραφο που θα αναφέρει τι θα προβλέπει η συνεργασία μας. Τέταρτη πτυχή, η κυρία Μογκερίνη θα το ε, θέσει στο Συμβούλιο τον Ιούνιο, θα παρουσιάσει θετικά την πρόσληψη των επιτετραμένων ασφαλείας όπως έχουν ε, κάτι αντίστοιχο η Γαλλία σε 8 χώρες μένα που επελέχθησαν θα προσελήφθησαν θα ξεκινήσουν το καλοκαίρι. Είναι σημαντικό για και τους λόγους αυτό, διότι πρέπει να έχουμε ανθρώπους με ιστορικό από δυνάμεις επιβολής του νόμου ή ε, μυστικές υπηρεσίες και όταν ξυπνάνε το πρωί να τους αρέσει να δουλεύουν στον τομέα και να αναπτύσσουν σχέση με τους ομολόγους τους. Δεύτερος λόγος, έχοντας ένα δίκτυο υπευθύνων που έχουν ασχοληθεί με τον τομέα μας βοηθά πάρα πολύ για να σχεδιάσουμε τη σωστή απάντηση και να έχουμε αποτελεσματικότερα προγράμματα δημιουργίας δυναμικού. Ε, πάμε στην πέμπτη πτυχή, συνεπώς πώς μπορούμε να βοηθήσουμε αυτές τις χώρες μαζί με τους συναδέλφους που έχουμε δραστηριοποιηθεί όλοι μαζί για να επισκεφτούμε τις διάφορες χώρες και για να εντοπίσουμε πού μπορούμε να τις βοηθήσουμε χρησιμοποιώντας το ISCSP, το πρώην ε, μέσο για την σταθερότητα και έχουμε δρομολογήσει αρκετά έργα και προγράμματα που θα ξεκινήσουν σύντομα, ένα στην Ιορδανία και καλωσορίζω την αντιπροσωπή από τη χώρα αυτή που είναι εδώ, 10 εκατομμύρια ευρώ είναι το πρόγραμμα της Ιορδανίας να βοηθήσουμε την Ιορδανία να επεξεργαστεί την πρόληψη, να αναπτύξει ένα όραμα, να εφαρμόσει, να υλοποιήσει το όραμα ε, κυρίως ε, να στηρίξουμε τους διάφορους φορείς κοινωνίας, 2,5 εκατομμύρια δίνουμε στο Λιβανό για να μειωθούν οι εντάσεις μεταξύ του τεράστιου αριθμού των προσφύγων. Ένας στους τρεις κατοίκους του Λιβάνου δεν είναι Λιβανέζος και προέρχεται από τη Συρία και να εργαστούμε τοπικά μέσα ενημέρωση στην τοπική αυτοδιοίκηση. Προσπαθούμε να βοηθήσουμε και την Εθνικό Σύμβουλο Ασφαλείας του Ιράκ να σχεδιάσει ε, μια άλλη προσέγγιση κατά πολέμηση τρομοκρατίας να σχεδιάσει και το Ιράκ μια προληπτική στρατηγική 3,5 εκατομμύρια πανέκη. Δεν θα σας προβληματίσω, θα σας αναφέρω τον κατάλογο, το λεπτομερή. Έχουμε ένα ειδικό πρόγραμμα το οποίο δημιουργήσαμε με την ΣΥΠΟΛ, την Υπηρεσία για την Κατάρτιση Αστυνομικών, διότι δεν έχουμε πρόγραμμα ε, επισκέψεων ανωτέρων ε, αξιωματούχων της ΜΕΝΑ στα Βαλκάνια θα θέλαμε λοιπόν να επισκέπτονται αυτοί οι αξιωματούχοι τους ομολόγους τους στην Ευρώπη, να ανταλλάσσουν εμπειρίες με τις διάφορες μονάδες τις ευρωπαϊκές και έχουμε διάφορα προγράμματα που θα εφαρμόσουμε με την ΜΕΝΑ στις χώρες Μαγκρέμπ. Πέμπτο, το έκτο. Είναι ένα θέμα που, όπου νομίζω ότι όντως έχουμε πρόοδο. Πρέπει να αναγνωρίσουμε βέβαια ότι δεν έχουμε κάνει τα πάντα, μένουν πολλά ακόμα να μάθουμε για να είμαστε πιο αποτελεσματικοί όσον αφορά την επικοινωνία μας. Η επικοινωνία είναι λοιπόν. Το πώς προβάλλεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, το πώς παρουσιάζει τη θέση της στον υπόλοιπο κόσμο είναι ένα ζήτημα. Γι' αυτό και είπατε εκπρόσωπος έχει μια ειδική task force για την επικοινωνία με συναδέλφους από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και με τη δικιά μου την ομάδα, ώστε να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε πώς μπορούμε να είμαστε περισσότερο παρόντες, να εξηγούμε καλύτερα το τι κάνουμε, να χρησιμοποιούμε τα κοινωνικά δίκτυα και να προβάλλουμε γενικά καλύτερα το έργο μας. Αυτό είναι το πρώτο βήμα. Δεν λέω ότι το έχουμε καταφέρει, αλλά είναι ένα βήμα που έχει γίνει προς τη σωστή κατεύθυνση. Το δεύτερο, που είναι της μόδας, αλλά και πολύ σημαντικό, πρέπει να βοηθούμε τις ίδιες τις χώρες να καταφέρουν να επικοινωνήσουν περισσότερο, να παρουσιάσουν καλύτερα αυτά που εκείνες κάνουν κατά της τρομοκρατίας, κατά του λεγόμενου Ισλαμικού κράτους, για παράδειγμα του Ντάς κλπ. Συμβουλεύουμε λοιπόν τις χώρες να έχουν τη δικιά τους στρατηγική επικοινωνίες. 12 από τις 24 χώρες μέχρι τώρα, το τελευταίο εξάμεινο, έχουν φτιάξει μια ομάδα περιγνωμόνων για να δούνε πώς θα προχωρήσουν επιτυχέστερα στην πολιτική τους επικοινωνίας. Γιατί άμα δείτε πόσο αποτελεσματικό είναι το λεγόμενο Ισλαμικό κράτος στη δικιά του την επικοινωνία, ε, αυτό σημαίνει ότι και εμείς πρέπει να είμαστε πολύ περισσότερο παρόντες στα κοινωνικά δίκτυα, στην επικοινωνία γενικά. Μια μελέτη που έγινε πρόσφατα δείχνει ότι έχει πάνω από 45.000 λογαριασμούς tweet το Ισλαμικό κράτος. Άρα πρέπει να δουλέψουμε όχι αφαιρώντας τα δικά τους, τις δικές τους σελίδες, αλλά παρουσιάζοντας καλύτερα τα δικά μας. Εδώ οι κυβερνήσεις έχουν να παίξουν το δικό τους ρόλο, αλλά πρέπει να βοηθήσουμε και την κοινωνία των πολιτών να το κάνει περισσότερο επίσης. Υπάρχει λοιπόν ένα πρόγραμμα πάνω στο οποίο δουλεύει η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης με εμπειρογνώμονες που θα τους διαθέσει περισσότερο. Και είναι κάτι που μας ζητιέται από όλες τις χώρες που επισκεπτόμαστε. Θέλουν τέτοιους εμπειρογνώμονες. Τώρα για την συμμαχία κατά του Ισλαμικού κράτους Κοίταξτε, επενδύουμε όλο και περισσότερες προσπάθειες ακριβώς στην ε, επικοινωνία μας αυτή. Το έβδομο θέμα είναι πώς θα κινητοποιήσουμε περισσότερο τους μηχανισμούς που έχουμε για την δικαιοσύνη στο εσωτερικό και προς τα έξω. Πώς δηλαδή τη Europol, τη Eurojust θα τις προβάλλουμε περισσότερο και τη CIPOL προς τα έξω. Για χρόνια οι χώρες μέλη διστάζανε, γιατί θεωρούσαν ότι οι υπηρεσίες αυτές έχουν φτιαχτεί κατεξοχήν και καταρχάς για να δημιουργήσουν τα δικά τους εσωτερικά δίκτυα και να λειτουργούν μέσα στις χώρες μέλη. Όμως ήρθε η ώρα, η Europol δημιουργήθηκε με τη συνθήκη του Μάστριχτ. Πάνε χρόνια. Ήρθε λοιπόν η ώρα να τους ζητήσουμε να δραστηριοποιηθούν περισσότερο και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης εξαιτίας των εξωτερικών απειλών ακριβώς. Με οικονομική στήριξη βέβαια πρέπει να προσαρμόσουν και το πρόγραμμα εργασίας τους, αλλά αυτό μπορεί να γίνει και στέλνοντας ε, στις χώρες που μας ενδιαφέρουν αξιωματούχους σύνδεσης. Liaison officers. Μπορούν να υπάρχουν και ειδικέ συμφωνίες συνεργασίας. Αν πάρω ένα παράδειγμα. Προσκαλούμε συστηματικά τους Τούρκους συναδέλφους σε συναντήσεις στη Eurojust, τακτικής. Προσπαθούμε να οργανώσουμε την πολιτική μας για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας στην Ευρώπη. Για αυτούς σημαίνουν πολλά αυτά, γιατί νιώθουν ότι ανήκουν και αυτοί στον ίδιο κύκλο. Αυτό θέλουμε να κάνουμε λοιπόν αλλά χρειάζεται χρόνος. Και θέλουμε να κάνουμε περισσότερα με την νομική βάση που διαθέτουμε. Μετά την 11η Σεπτεμβρίου εγώ είχα φέρει την ιδέα για ενισχυμένη συμφωνία και έκδοσης και νομική συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Εξυγχρονίσαμε λοιπόν με διαπραγματεύσεις και για τις 28 χώρες μέλη και έχουμε τώρα ενιαίες συμφωνίες έκδοσης με τις ΗΠΑ για να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις του 21ου αιώνα. Το ίδιο θέλουμε να κάνουμε και με τις χώρες γύρω από τη Μεσόγειο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δηλαδή να διαπραγματευτεί εκ μέρους των 28 χωρών. Όταν έχουμε ένα κέντρο αριστείας θα ήταν καλό οι εμπειρογνώμονε των χωρών μελών να είναι διαθέσιμοι για να βοηθούν τις χώρες γύρω από τη Μεσόγειο. Με δύο λόγια, αυτά προσπαθούμε να κάνουμε. Και τέλος, τέλος, πριν από λίγους μήνες δημιούργησα μία ομάδα εμπειρογνωμόνων για τους ξένους μαχητές από χώρες, από το Μαρόκο μέχρι την Τουρκία. Συναντηθήκαμε και στις Βρυξέλλες και στο Ραμπάτ και μας προσκάλεσαν να πάμε κι αλλού για την τρίτη συνάντηση στη Βαγδάτη. Είναι σημαντικό γιατί σήμερα έχουμε περισσότερες πληροφορίες, τι μοιραζόμαστε μεταξύ μας και προσπαθούμε από κοινού να βρούμε μια απάντηση. Και το τελευταίο τελευταίο, μετά θα σταματήσω. Άλλες προκλήσεις. Χρειαζόμαστε οικονομικούς πόρους. Αν θέλουμε να βοηθήσουμε περισσότερο και να έχουμε περισσότερη πραγματογνωμοσύνη στη διάθεσή σας, πρέπει να αυξηθεί και το κονδύλι για τον αντιτρομοκρατικό αγώνα. Να υπάρχει ο στόχος, όπως τώρα στο σημερινό δημοσιονομικό πρόγραμμα. Δεύτερον, να έχουμε εμπειρογνώμονες διαθέσιμους από τις χώρες μέλη. Όπως καταλαβαίνετε, το Υπουργείο Εσωτερικών θέλει να τους κρατάει στις χώρες. Παρ' όλα αυτά πρέπει να είναι ε, διαθέσιμοι για να πάνε δύο μήνες για παράδειγμα στη Βαγδάτη. Έπειτα, υπάρχει το θέμα του κινδύνου. Όταν κάποιος δουλεύει για να αντιμετωπίσει την τρομοκρατία, υπάρχει ο κίνδυνος και της αποτυχίας. Μερικές φορές είμαστε αντιμέτωποι και με συγκεκριμένα συμφέροντα. Βλέπετε, υπάρχουν δυνάμεις μέσα στις χώρες καμιά φορά που χρειάζονται μεταρρύθμιση. Τέλος, διμερείς σχέσεις και πολυμερείς σχέσεις. Εδώ πρέπει να βρεθεί το σωστό μείγμα, γιατί υπάρχουν πολλά, όπως το φόρουμ κατά της τρομοκρατίας, από η Χίλαρη Κλίντον πριν από χρόνια. Υπάρχουν τα Ηνωμένα Έθνη, υπάρχουν ε, η Ιντερπολ, διάφορα δηλαδή πολυμερή μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας. Αλλά πρέπει όλα αυτά να τα συνδυάζουμε με τη σωστή πάντα με διμερείς σχέσεις. Η ένταση των σχέσεων αυτών εξαρτάται από το ιστορικό, από τις ειδικέ σχέσεις που έχουμε με μερικές χώρες και αυτές τις σχέσεις πρέπει να τις αναπτύσσουμε όλοι μαζί. Αυτά είχα να πω. Ευχαριστώ πολύ και ελπίζω έτσι να σας έδωσα αρκετές πληροφορίες. Ο Πρόεδρος Πάσκου σας ευχαριστώ πολύ. Πριν να αρχίσουμε τώρα την συζήτηση με τους συναδέλφους, να απευθύνω χαιρετισμό εδώ στην αντιπροσωπεία της συνελεύσεως του Βασιλείου της Ιορδανίας. Και αν δεν κάνω λάθος, ο επικεφαλής της αντιπροσωπείας είναι ο κύριος Σουλεϊμάν Αλζαμπέν που είναι και ε, αντιπρόεδρος της συνελεύσεως. Είναι ορθό αυτό, μάλιστα, ενεύουν καταφετικά οι προσκεκλημένοι και παρακολουθούν την συζήτησή μας τα πρόσωπα αυτά. Καλώς ήρθατε λοιπόν. Θα παρακαλέσω τώρα τον κύριο Τάνοκ, ο οποίος είναι εισηγητής της Επιτροπής Εξωτερικών για την γνωμοδότηση, για την έκθεση, για την αποτροπή η πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησεως για την έκθεση κυρία Ντάτη δηλαδή. Πολύ σύντομα κύριε Πρόεδρε, λέει ο κύριος Τάνοκ και βεβαίως ένα θερμό καλώς ορίσατε στον ε, προσκεκλημένο μας ε, είστε έμπειρος πλέον για τα θέματα αυτά Νομίζω πράγματι μας δώσατε μια ευρεία επισκόπηση των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν 28 χώρες μέλη και μεμονωμένα αλλά και συλλογικά στον αγώνα που διεξάγουμε κατά τη διεθνούς Δημοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος και υπέρ της ασφαλείας των πολιτών μας. Θα ήθελα να πιστεύω ότι πιο μακροπρόθεσμα και για μια χώρα όπως η δική μου, το Ενωμένο Βασίλειο δηλαδή, όπου υπάρχουν πάνω από χίλιες, χίλιες τζιχαντιστές οι οποίοι πολεμούν στις τάξεις του ISIS του Ισλαμικού κράτους στην ε, Συρία και στο Ιράκ. Θα θέλαμε μια πιο μακροπρόθεσμη στρατηγική πρόληψη. Έχουν γίνει προσπάθειες από την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου. Είναι δύσκολο να εντοπιστούν οι νέοι αυτοί νέοι άντρε σε ένα πρώιμο στάδιο γιατί ριζοσπαστικοποιούνται και προχωρούν να στρατολογούν πρόσωπα για να γίνουν αυτά μαχητές ε, του ISIS. Αυτά είναι και δαπανηρά, δηλαδή χρειάζεται και κονδύλια και προσωπικό με ιδιαίτερη εμπειρογνωμοσύνη. Κατά τη γνώμη μου αυτό που χρειάζεται είναι να κοιτάξουμε ποιες είναι οι καλύτερες πρακτικές οι οποίοι υπέρ των οποίων συνηγορούν και οι περισσότερες χώρε μέλη. Η Γερμανία ηγείται τι προσπάθειε αυτής από πολλές απόψεις. Θα πρέπει να δούμε και τι γίνεται και στο εθνικό επίπεδο και εκεί η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να συλλέξει τα δεδομένα, να συλλέξει τις ενδείξει και να παίξει και ένα ρόλο καθοδηγητικό. Έχω όμω και ορισμένε ερωτήσει για Προ λίγων εβδομάδων εμφανίστηκε στον τύπο είδηση ότι συνελήφθη ύποπτο στην Ιταλία που θεωρήθηκε ότι ήταν παρόν στην τρομοκρατική επίθεση στο Μουσείο της Τινησίας και ότι αυτός ο άνθρωπος ζούσε στην Ιταλία ως πρόσφυγας. Είχε ίσως μάλιστα περάσει και με μία από τις γνωστές αυτές βάρκες την Μεσόγειο. Υπάρχει κατά τη γνώμη σας σημαντικός κίνδυνος διείσδυσης μεγάλων, μεταξύ των μεγάλων αριθμών προσφύγων που περνούν την θάλασσα με, ε, ασφα, με ανασφαλή σκάφη να διεισδύσουν και τρομοκράτες. Επίσης μιλήσατε στην παρέμβασή σας για την Ιντερπολ και για το ενδεχόμενο να συμβάλλει στον αγώνα αυτό. Πώς απαντάτε σε εκείνους που λένε ότι καμιά φορά η Ιντερπολ και ορισμένες χώρες μέλη καταχρώνται το σύστημα της ΕΛΘΑΣ κάρτας. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Φωτίγκα, που είναι η πρόεδρος της Υποεπιτροπής Ασφάλειας και Άμυνας. Ευχαριστώ. Καλώς ήρθατε κύριε Κέρκχοφ στην Ευρωβουλή. Σας ευχαριστώ και για την παρέμβασή σας. Με ικανοποιεί ιδιαίτερως η δηλώσει σα σχετικά με τις προσπάθειες που καταβάλλετε για να αντιμετωπίσετε την προπαγάνδα του Ισλαμικού κράτους και άλλων εξτρεμιστικών ομάδων ε, που προσπαθούν να επηρεάσουν την κοινή γνώμη στις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης μεταξύ άλλων. Χαίρομαι και για την συντονισμένη δράση για την πρόσληψη συμβούλων για την διατήρηση των στρατηγικών επικοινωνιών. Η ερώτησή μου έχει σχέση, μάλλον ζητώ να μάθω ποια είναι η εκτίμησή σας σχετικά με τον συντονισμό κατά του της προ, προσπάθειας που κάνει η ISIS με παραπλάνηση και με άλλα μέσα. Τι είδους αντίδραση χρειάζεται. Και όπως συζητήσαμε και την συνεργασία με τρίτα μέρη ή τρίτες χώρες, τρεις επικεφαλίδες, Ρωσία, Τουρκία και Ιράν. Μετά από τις αποφάσεις του Μετβιέντεφ για το Αφγανιστάν, τι έχετε να πείτε γι' αυτό, για το Ιράν, μπορούμε να αναμένουμε συνεργασία με την χώρα αυτή. για την στήριξη μειωνοτικών ομάδων μέσα στην, ε, στο Ιράκ όπως τους Γεζίδης για παράδειγμα και η Τουρκία είναι άλλο βέβαια θέμα ιδιαίτερα ευρύ. Ε, τώρα έχουμε κλείσει τον κατάλογο. Δεύτερο θα ήθελα να παρακαλέσω όλες και όλους να τοποθετήσετε μέσα σε ένα λεπτό. Γιατί είναι παρόν και ο κύριος Μπρόκ που θα αναλάβει στις 6. Κύριε Πρέκοβιτς, έχετε τον λόγο. Για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Δεκερχόβε. ευχαριστώ που ήρθατε και μάλιστα τόσο σύντομα πάλι στην Επιτροπή Εξωτερικών. Δείχνει βεβαίως αυτό και τη σημασία του θέματος το οποίο συντονίζεται εδώ και μια δεκαετία. Έχετε ανταλλαγή δεδομένων με χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Έχουμε περίπου 600 ανθρώπους από χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης προς ε, Μέση Ανατολή, κυρίως από Βοσνία, Ζουγοβίνη, Κόσοβο, ε, Μακεδονία. Πού βρίσκονται οι ανταλλαγές δεδομένων ε, που έχετε προχωρήσει, σε έχετε προχωρήσει. Η κυρία Γκόμες, 1,5 λεπτό. Καλώς ήρθατε και Ντεκερκόβε. Πώς αξιολογείτε την ανταλλαγή πληροφοριών. Έχει βελτιωθεί μεταξύ χωρών μελών και των οργανισμών όπως της Ευρωπόλ για το λαθρεμπόριο όπλων. Είπατε ότι θα ε, καταθέσει νέα πρόταση κανονισμού η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μα υπάρχει κοινή θέση του Συμβουλίου. Αρκεί να την εφαρμόσουν την κοινή θέση οι χώρε μέλη. Θα κολλήσουμε τώρα με την επεξεργασία του νέου κανονισμού και παραμελώντας την κοινή θέση που ήδη υπάρχει. Εγώ είμαι μεταξύ εκείνων που απορρίπτω την ιδέα να βάλουμε όλους το ίδιο καλάθι τρομοκράτες και πρόσφυγες Όπω προσπαθούν ορισμένοι να πράξουν για να φοβήσουν την κοινή γνώμη. Γνωρίζω βέβαια ποια είναι η κατάσταση στην Λιβύη, η οποία Λιβύη είναι τώρα ασφαλής λιμίν για του τρομοκράτε. Ποιε είναι οι πληροφορίε που διαθέτεται, γιατί βεβαίω ο στόχο του δεν είναι η ίδια η Λιβύη, είναι η Ευρώπη. Ποιε πληροφορίε μπορείτε να μα δώσετε σχετικά. Και τέλο, οι χώρε μέλη μα συντονίζονται καλύτερα στη γραμμή αυτή του μετόπου που είναι το Ιράκ απέναντι στους τρομοκράτες του Ισλαμικού κράτους. Μιλήσατε και για τον συντονισμό με την Τουρκία για το ΠΚΚ. Αυτό επεκτείνεται και στον Άισις και στην Σαουδική Αραβία και στο Κατά. Ευχαριστώ κύριε Στεμές Μάκερ. Ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. Καλώς ήρθατε κύριε Τεκερκόφερ. Δύο σύντομες ερωτήσεις έχω παρακαλώ. Μετά την τρομοκρατική επίθεση στο Παρίσι, έλαβαν χώρα διάφορες δράσεις στη Γαλλία και στην Ολλανδία, ε, κρατήσεις, συλλήψεις και τσετσένων που είχαν ρωσικό διαβατήριο. Στο Βερβιέ, στο Βέλγιο επίσης κάποιος τσετσένος έχασε τη ζωή του. Τι φαίνεται υπήρχαν όπλα από τη Βοσνία. Ο παράγοντας ε, Τσετσένοι φαίνεται ότι παίζουν ρόλο και στην σύγκρουση στην Ουκρανία. Οπότε δεν θα έπρεπε να συμπεριλάβουμε και την κυβέρνηση της Ουκρανίας στη συνεργασία στην Ευρώπη κατά της τρομοκρατίας. Δεύτερον, 22 Απριλίου στο Μπαχρέιν, στο Συμβούλιο για τη Συνεργασία των Χωρών του Κόλπου έγινε ένα εργαστήριο όσον αφορά τη χρηματοδότηση του λεγόμενου Ισλαμικού κράτους από τις χώρες του Κόλπου και την Ευρώπη. Ξέρετε τι συζητήθηκε εκεί και μεταφέρθηκαν οι ανησυχίες της Ευρώπης για το ρόλο της Σαουδικής Αραβίας και του κατάστη χρηματοδότηση του Ισλαμικού λεγόμενου αυτού κράτους. Και υποσχέθηκε το Συμβούλιο αυτό να κάνει κάποιες προσπάθειες. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Κύριος Κόζου. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Λέω κύριο Σκούζο. Όσον αφορά το PNR, τα στοιχεία των επιβατών Νομίζω ότι δεν μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει την επίθεση στο Τσάρλι Εμπδό για να πουλήσουμε εμείς αυτά τα στοιχεία. Όχι, ξέρουμε πολύ καλά ότι δύο τουλάχιστον μυστικές ευρωπαϊκές υπηρεσίες παρακολουθούσαν τους δράστες, τους γνωρίζανε. Έτσι λοιπόν, με την αίσθηση που δημιουργείται από μια τέτοια τρομοκρατική επίθεση, στη συνέχεια προσπαθούμε να περιορίσουμε τις ελευθερίες των πολιτών. Είδα από το 2013. Μα πώς χρησιμοποιούνται τελικά τα δεδομένα των Ευρωπαίων. Ξέρουμε ότι η NSA έκανε την μεγαλύτερη κατασκοπική δράση. Όμως οι Ηνωμένε Πολιτείες μεν αποφάσισαν να διακόψουν κάποια από τα προβλήματα, κάποια από τις δράσεις αυτές, όχι όμως και το Ηνωμένο Βασίλειο. Εγώ δεν έχω ακούσει τίποτα πέρα από το ότι χρησιμοποιείται η τρομοκρατική αυτή επίθεση για να πουλήσουμε τα PNR. Όμως, οι πολίτες μας πρέπει να καθησυχαστούν ότι δεν θα χρησιμοποιηθούν τα δεδομένα τους, ότι δεν θα τους κατασκοπεύουμε. Ευχαριστούμε. Η κυρία Λόχμπίλερ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Κερχόφε για την πολύ ενδιαφέρουσα ομιλία σας. Έχω μία-δύο ερωτήσεις που έχω να σας θέσω. Πρώτα απ' όλα με ενδιαφέρει η χρήση των μη επανδρομένων οχημάτων, drones, στις αντιδρομοκρατικές επιχειρήσεις. Ακούσαμε από τη ΣΥΠΑ ότι έχουν σκοτωθεί και πολίτες με τα οπλισμένα αυτά μη επανδρομένα ε, οχήματα όπως ο Τζοβάνι Λαπόρτο. Ε, ελήφθησαν κάποια μέτρα σχετικά με την Αμερικανική κυβέρνηση που χρησιμοποιεί τα drones. Ποια είναι η θέση σας όσον αφορά την χρησι... αυτών των οπλισμένων ε, μη επανδρομένων οχημάτων στην καταπολέμηση τρομοκρατίας του Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 2014 είχαμε ψηφίσει ψήφισμα, ψήφισμα με το οποίο ζητούσαμε συγκεκριμένο νομοθετικό πλαίσιο για την χρήση των μη επανδρομένων αεροσκαφών. Τι γνώμη έχετε. Τώρα, βλέπουμε ειδήσει κυρίως από την Βόρεια Αφρική ότι οι χώρες μέλη προτίθενται να δημιουργήσουν βάσεις μη επανδρομένων αεροσκαφών στο Μαρόκο και στην Τινησία. Έχετε σχετικές πληροφορίες και Υπάρχει και ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ του Αραβικού Συνδέσμου και του EIS σε θέματα αντιτρομοκρατίας. Είναι μέρος αυτής της ενισχυμένης συνεργασίας αυτή η μετακίνηση βάσεων μη επανδομένων ασκαφών στην Βόρεια Αφρική. Ο κ. Κάρβερ, σας παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Τεκερκόφ. Ανησυχείτε για στην ασφάλεια εκείνων που εργάζονται και τη δημοκρατία και κυρίως μετά από αυτά που συνέβησαν με την αποκαλύψη Σνόντερ. Πώς θα γίνεται το μοίρασμα των πληροφοριών μεταξύ των μελών και η καλύτερη συνεργασία με τις μυστικές υπηρεσίες Τουρκίας. Αναφερθήκατε σε κάποια πρόσκληση να παραστούν στις συνεδριάσεις του Eurojust για την τακτική. Αυτό ε, σύγχρονα με το οποίο ε, στέλνουν στους επαναστάτες του Ισλαμικού κράτους στη Συρία ε, οι μυστικές υπηρεσίες Τουρκίας. Τι γίνεται με τη, τι γίνεται με τη δίσδυση ενδεχομένω μαχητών στην Ευρώπη μέσω των προσφύγων που έρχονται εδώ λόγω της ε, κρίσης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, κύριε Ντεχέρχοφ, θα ήθελα και εγώ ε, να σας κάνω μια ερώτηση σχετικά με το PNR, τα στοιχεία τα οποία συλλέγουμε, όπως είπατε, σε συνεργασία με τους φίλους μας τους Αμερικανούς για τους ταξιδιώτες πώς θα εξασφαλίσουμε ότι τα στοιχεία αυτά δεν θα χρησιμοποιηθούν για εις βάρος πιθανών πολιτικών αντιπάλων, τους οποίους θα μπορούσαμε να κατηγορήσουμε ως πιθανούς τρομοκράτες και με τον τρόπο αυτό να προσπαθήσουμε να τους ε, εξοβελήσουμε από την πολιτική σκηνή μιας χώρας. Στη χώρα μου δυστυχώς στην Ελλάδα έχουμε τέτοιες περιπτώσεις. Και η δεύτερη ερώτηση είναι η εξή. Είπατε ότι η προσπάθεια για την αντιμετώπιση του αντισημιτισμού και του, της Ισλαμοφοβίας θα συμβάλλει στην αντιμετώπιση της τρομοκρατίας. Θα ήθελα σας παρακαλώ να μου αναλύσετε αυτή τη θέση, πώς δηλαδή αυτή η προσπάθεια θα συμβάλλει στο να αντιμετωπίσουμε την μορφή της ε, τρομοκρατίας που αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή, η οποία κυρίως προέρχεται από Ισλαμιστές. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ, ο κύριος Γιούρεκ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Ντεκέρκοφ. Θα ήθελα επίσης να σας ρωτήσω αν μπορείτε να μου πείτε το εξής. Το πρώτο που μας προβληματίζει είναι η κλίμακα της εκροής τζιχαντιστών, μαχητών από την Ευρώπη. Τι είναι αυτό το φαινόμενο, κοινωνιολογικό, κοινωνιολογικό φαινόμενο που ε, ε, εστιάζεται στις κοινότητες στις οποίες ανήκουν ή οφείλεται σε εκστρατεία που έχει σαν στόχο την νεολαία της Ευρώπης. Έχουμε πληροφορίες που χρονολογούνται εδώ και μερικούς μήνες αυξάνεται αυτή η εκροή των ξένων πολεμιστών, των Ευρωπαίων πάνω πολεμιστών στο πλευρό του Ισλαμικού κράτους ή όχι. Ποιος οργανώνει αυτή, αυτή τη στρατολόγηση. Ακτιβιστές της ISIS ή υπάρχουν μόνιμα δίκτυα στην Ευρώπη που κάνουν αυτή τη δουλειά. Μετά αναφερθήκατε σε προληπτικά μέτρα που θα πρέπει να εφαρμόζονται όσον αφορά τους τζιχαντιστές που επιστρέφουν από τις αραβικές χώρες. Ξέρουμε πώς συμπεριφέρονται αυτοί μετά αφού επιστέψουν στην Ευρώπη. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μπασίρ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δίνετε αυτή την ευκαιρία. Θα ήθελα να πω ότι θλίβομαι λέγοντας ότι οι προσπάθειές σας θα πετύχουν ελάχιστα. Κατά την άποψή μου είναι σαν να προσπαθούμε να βάλουμε τον δόκρεμα ξανά στο σωληνάριο αφού έχει βγει σαν να προσπαθήσουμε να ξανακολλήσουμε ένα βάζο μίγκα αφού έχει ε, Αυτά που κάναμε στη Μέση Ανατολή με ε, στη Μέση Ανατολή αυτό που κάναμε στη Γερμανία με το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο να έχουμε ένα σχέδιο Μάρσαλ εάν δεν το είχαμε κάνει αυτό στη Γερμανία η Γερμανία θα μπορούσε να είναι ένα χρεοκοπημένο κράτος μήπως χρειάζεται να κάνουμε αυτό εδώ αν δείτε χώρες όπως είναι το Αφγανιστάν, η Λιβύη, το Ιράκ, η Συρία βλέπουμε ότι δεν υπάρχει κεντρική κυβέρνηση, δεν υπάρχει αστυνομία, δεν υπάρχει στρατός για να ελέγχουν τους εξτρεμιστές, τους τρομοκράτες. Αυτό που χρειάζεται να κάνουμε είναι να τους βοηθήσουμε. Δείτε τι γίνεται στο Πακιστάν πέρσι. Επειδή υπήρχε στρατός, επειδή υπήρχε αστυνομία, έφεραν τον πόλεμο στους τρομοκράτες και ε, υποχωρούν οι Ταλιμπάν και κερδίζει το κράτος. Αν δεν ενισχύσετε το κράτος, τότε θα αποτύχουμε. Είμαστε καταδικασμένοι σε αποτυχία. Επικροτώ τις προσπάθειές σας. Πρέπει να συνεχιστούν οι προσπάθειες, αλλά όλες αυτές οι προσπάθειες, αν δεν τα κάνουμε αυτά, θα αποτύχουν. Ευχαριστώ. Κύριε Ντεκέρκοφ, σε αυτή την θετική νότα μπορείτε να αρχίσετε τις απαντήσεις σας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ για τις δύσκολες ερωτήσεις σας. Με τη σειρά θα προσπαθήσω να απαντήσω. Για τον κίνδυνο. Κίνδυνο δίσδυσης τρομοκρατών στο κύκλωμα των ε, μεταναστών Όντω πρέπει να υπάρχει πάντα διάκριση ανάμεσα στους μετανάστες και τους εγκληματίες. Έχω χρόνια εδώ. Οι στόχοι τους είναι διαφορετικοί. Οι μετανάστες θέλουν μια διαφορετική ζωή, μια καλύτερη ζωή. Υπάρχουν και εκείνοι που χρήζουν διεθνούς προστασίες. Ε, οι τρομοκράτες είναι κάτι διαφορετικό βέβαια. Από αυτό που γνωρίζω από το τι γίνεται στη Λιβύη, όντως το λεγόμενο Ισλαμικό κράτος, το ISIS, φαίνεται ότι εμπλέκεται στη, στο λαθρεμπόριο ανθρώπων, ουσιαστικά από εκεί έχουν και μέρος των κερδών τους. 5.000 πρέπει να πληρώνει ο καθένας από ό,τι έχω καταλάβει. Δεν ξέρω αν χρησιμοποιούν το δίκτυο ήδη, οι για να μπαίνουν στην Ευρώπη. Εγώ νομίζω ότι προς το παρόν, όπως είπε και κάποιος εδώ, Κυρίως πρόκειται για μαχητές Ευρωπαίους που πηγαίνουν εκεί να πολεμήσουν. Δεν χρειάζονται το δίκτυο των παράνομων μεταναστών, γιατί αυτοί θα χρειαζόντουσαν κάποιο διαβατήριο. Το οποίο είναι αρκετή το χρειαζόμαστε. Το χρειαζόμαστε γιατί ορισμένοι ακριβώ πηγαίνουν με το αεροπλάνο και δεν είναι γνωστοί ούτε από τι μυστικέ υπηρεσίε ούτε από την αστυνομία και μπορούν να φύγουν και να πάνε στη Συρία λέγοντας ότι πάνε διακοπές στην Τουρκία καταρχήν. Δεν νομίζω δηλαδή ότι το ISIS χρειάζεται ε, να δυσδύσει στο δίκτυο μεταναστών για να κάνει τη δουλειά του. Βέβαια, βέβαια, παρόλα αυτά, σίγουρα πρέπει να πιέσουμε περισσότερο την Frontex στην αντιμετώπιση εγκλημάτων για ιστορικούς λόγους κι άλλους. Τη Frontex τη φτιάξαμε σε αυτό που πριν λέγαμε ε, Η Frontex δηλαδή έχει ως αποστολή και την καταπολέμηση του εγκλήματος, αλλά την μεταναστευτική ροή. Όμως τελικά ο συνοριοφύλακας αναγκαστικά θα έρθει αντιμέτωπος και με εγκληματίες. Τώρα δεν έχουμε τους πυλώνες πρώτος, δεύτερο τρίτος με τη συνθήκη της Λισαβόνας, ακόμα και αν η ΚΕΠΑ είναι κάτι διαφορετικό. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε λοιπόν την κοινοτική μέθοδο. Και αν έπρεπε σήμερα να κάνουμε τη Frontex, η Frontex θα αναλάμβανε και τη συλλογή προσωπικών δεδομένων βάσει κάποιων κανόνων σε συνεργασία με το Europol. Και εγώ θέλω η Frontex και η Europol να έχουν όσο γίνεται πιο γρήγορα μια λειτουργική συνεργασία, επιχειρησιακή συνεργασία γιατί είναι κάτι που χρειαζόμαστε όταν έχουμε μια κοινή δράση στη Μεσόγειο και συλλέγονται ονόματα ανθρώπων που σώζουμε στη θάλασσα και λένε ότι ξέρουν κάποιον που είναι στην Κωνσταντινούπολη και αυτός είναι επικεφαλής ενός δικτύου, ε, τότε θα έπρεπε να ζητήσουμε από την Κυρούπολη να ψάξει τα διάφορα, τις διάφορες βάσεις δεδομένων που έχει και έτσι θα αποφεύγαμε με την εμπορία αυτή ανθρώπων, την παράνομη μεταφορά τους να κερδίζουν εκατομμύρια και εκατομμύρια αυτοί οι εγκληματίες. Δεύτερον, Ίντερπολ. Ο κύριος Τάνοκ ρώτησε. Οι χώρες μέλη είναι πολύ προσεκτικές όταν χρησιμοποιούν την Ιντερπολ να μην ε, πηγαίνουν ευαίσθητες πληροφορίες σε όλες τις χώρες της Ιντερπόλ. Ότι κάποιες μπορεί να χρησιμοποιήσουν διαφορετικούς τρόπους. Πρέπει, αν υπάρχουν λόγοι ευαίσθητοι και φοβούμαστε ότι θα χρησιμοποιηθούν για πολιτικούς λόγους, τότε να μην περνάνε στο σύστημα έτσι απρόσκοπτα. για περισσότερη συνεργασία με τη Ρωσία, την Τουρκία και το Ιράν. Συμφωνώ. Και ελπίζω όταν θα τελειώσουν οι διαπραγματεύσεις μας για το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα με το Ιράν, ελπίζω τη σχέση αυτή να μπορέσουμε να τη χρησιμοποιήσουμε περισσότερο. Η Ρωσία είναι ένα θέμα Μάλλον με τη Ρωσία έχουμε κάποιες συγκλήσεις απόψεων για την καταπολέμηση της Αλκαΐντα. Και βέβαια η Τουρκία είναι ένας πολύ στενός εταίρος. Αυτό που ρωτήσατε εσείς για τα Βαλκάνια. Δεν είμαι σε θέση να σας απαντήσω τώρα, γιατί δεν μπορώ να ελέγξω τις πληροφορίες εγώ ίδιος. Αλλά όταν πάω στα Βαλκάνια και θα πάω γιατί θέλουμε περισσότερη συνεργασία μαζί τους για την καταπολέμηση των ε, ξένων μαχητών, είπατε 700 μπορεί να και παραπάνω. Εντυπωσιάστηκα και στο Κωσοϊβοπέδιο και στη Βοσνία Ζεγοβίνα και στη Σερβία εντυπωσιάστηκα από τους συνομιλητές μου. Είναι νέοι αξιωματούχοι και εντυπωσιάστηκα γιατί συνεργάζονται πολύ και μεταξύ τους και πολύ καλά. Αλλά δεν είμαι σε θέση να σας απαντήσω για την ποιότητα των πληροφοριών αυτών καθ' αυτών. Και να απαντήσω στην Άννα Γκόμες για τον επιβεσμό των πληροφοριών. Αύριο θα πάω στο Συμβούλιο λέγαμε μέχρι τώρα για τις πληροφορίε που δίνουμε στη Europol και στη Eurojust. Είναι αλήθεια ότι όλο και περισσότερα δεδομένα μοιραζόμαστε μαζί τους. Για το λαθρεμπόριο όπλων, οι χώρες μέλη έχουν διαφορετικές εντολές όταν πρόκειται για τον αφοπλισμό. Και σε μερικές περιπτώσεις είναι πολύ εύκολο αφού παροπλήσετε ένα όπλο μετά να το ξαναχρησιμοποιήσετε. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει οι προδιαγραφές να είναι υψηλότερε δυνατόν. Και θα ζητήσω ρύθμιση, όχι οδηγία, γιατί η οδηγία θα πάρει χρόνια. Κύριε Ντεμασμάκερ, ρωτήσατε για την Ουκρανία. Είναι ένα λεπτό θέμα. το κατά πόσο υπάρχουν, δεν υπάρχουν μαχητές. Όντως κάποιοι Ευρωπαίοι έχουν πάει στην Ουκρανία. Έχουμε ζητήσει συνάντηση με τις υπηρεσίες πληροφοριών να συνεργαστούμε στο θέμα της αντιτρομοκρατίας. Σε δύο εβδομάδες νομίζω θα πάω εκεί και εκεί θα μιλήσω μαζί τους και θα δούμε πώς μπορούμε να τους βοηθήσουμε. Κύριε Κουζό, το PNR. Λέτε δεν θα είχε αποφύγει την επίθεση στο Παρίσι. Μα νομίζω ότι κανένας δεν ε, είπε ότι αν είχαμε το PNR θα είχαμε εμποδίσει την τρομοκρατική αυτή επίθεση στο Σαρλί επτό. Εξάλλου, μήνες πριν το Παρίσι εγώ πίεζα για το PNR. Θα ήταν άδικο δηλαδή να χρησιμοποιήσουμε το Παρίσι σαν δικαιολογία για το PNR, είτε προς τη μία κατεύθυνση είτε προς την άλλη κατεύθυνση όμως. Να είμαστε ειλικρινεί. Και εγώ πάντα λέω ότι το χρειαζόμαστε το PNR, όχι επειδή έγινε τρομοκρατική επίθεση στο Σαρλί Επδό, αλλά γιατί είναι ο μόνος τρόπος να εντοπίσουμε επικίνδυνους ε, ε, επισκέπτες μας. Για τα drones τώρα, τα μη πανδρομένα αεροσκάφη. Θα είμαι απλοϊκός. Θυμάμαι. Πέρυσι στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για την Άμυνα η εξωτερική υπηρεσία, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικών Σχέσεων άρχισε να δουλεύει πάνω σε αυτό το θέμα. Δεν υπήρχε επίσημη θέση της Ευρώπης. Μα αυτό που διακυδεύεται εδώ δεν είναι το drone, δεν έχει καμιά διαφορά με το jet fighter, δεν είναι δηλαδή το μέσον το πρόβλημα. Το θέμα είναι πώς χρησιμοποιείται, αν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για επίθεση. Στα πλαίσια λοιπόν συγκρούσεων είναι που συζητιέται με τους Αμερικανούς. Και από τον πρώτο μπούς είχαμε την στάση των Αμερικανών για την αποτροπή. Αρχίσαμε τότε με το νομικό σύμβουλο του State Department τη συζήτηση, συνεχίσαμε και την ερμηνεία που δίνουν εκείνοι για τον ε, νόμο για την αντιμετώπιση πολεμικών πράξεων ή τρομοκρατίας. Δεν γνωρίζω να υπάρχει συμφωνία για την Ισία, Αλγερία και λοιπά να χρησιμοποιηθούν ως στρατιωτική βάση για drones. Και δεν νομίζω ότι οι Ευρωπαίοι τα βλέπουν όπως τα βλέπουν οι Αμερικανοί. Έχουμε κάποια drones για παρατηρήσεις, αλλά όχι για επιθέσεις. Στην Ιγυρία ξέρω ότι υπάρχει μόνο μια ε, βάση των Αμερικανών όμως. Για όπλα προς τη Συρία δεν ε, το γνωρίζω. Έχω καλές σχέσεις με τα ΜΕΤΗ και κάθε φορά που πηγαίνω στην Τουρκία συναντιέμαι με τον κύριο Κουφιντάν είναι υπηρεσία που μας δίνει πολλές πληροφορίες για τη Συρία. Για την Ισλαμοφοβία και τον αντισημιτισμό και την τρομοκρατία, δεν λέω ότι υπάρχει άμεση σχέση. αυτή η διαδικασία της ζωστικοποίηση, ο ρατσισμός είναι ίσως ένα στοιχείο που μπορεί να οδηγήσει κάποιους να πέσουν στην βία. Δεν είναι όμως ο μόνος παράγοντας και δεν είναι και άμεση σχέση. Τα στοιχεία που ξέρουμε από τη Γαλλία είναι ενισχυτικά και δείχνουν ότι υπάρχει κάποια άνοδος του αντισημιτισμού. Το ξέρω και από το Βέλγιο. 7.000 έφυγαν πέρυσι και θα φύγουν περισσότεροι φέτος από ό,τι φαίνεται. Και το είπε και ο Πρωθυπουργό μετά την επίθεση στο Σαρλί Επντό. Έγιναν επιθέσεις εναντίον Εβραίων επειδή ήταν Εβραίοι. Και αυτό είναι παράδεκτο. Ξέρω ότι στη Γαλλία γίνεται η συζήτηση για το κατά πόσο η λέξη Ισλαμοφοβία πρέπει να μπει στο ίδιο επίπεδο με τον αντισημιτισμό. Είναι κάτι διαφορετικό, γιατί η επίθεση, ο αντισημιτισμός έχει να κάνει με την επίθεση κατά των Εβραίων επειδή είναι Εβραίοι. Όχι επειδή είναι άνθρωποι που ακολουθούν ε, έντονα την θρησκεία τους, ενώ ε, στην περίπτωση της Ισλαμοφοβίας είναι διαφορετικά τα πράγματα. Και η επίθεση στο μουσείο στην ε, Ισία το έδειξε. Γίνονται επιθέσεις Ισλαμιστών και κατά Πρέπει λοιπόν να αποφύγουμε τη ζωστικοποίηση, αυτό είναι σίγουρο. Και ευχαριστώ πολύ τον Αντιπρόεδρο Τίμερμανς για τα όσα κάνει γι' αυτό. Για τους ξένους μαχητές, και εδώ βέβαια θα χρειαζόμασταν περισσότερο χρόνο να εξηγήσουμε ποια είναι η διαδικασία πρόσληψης, ριζαστικοποίησης των ανθρώπων αυτών. Τα κοινωνικά δίκτυα σίγουρα παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο. Στο Βέλγιο το Βέλγιο έχουμε τους περισσότερους που φεύγουν για τη Συρία και το Ιράκ. Γιατί, γιατί έχουμε ε, εδώ πέρα τη Σαριά for Belgium που είναι μια οργάνωση σελαφιστών ενεργός. Οι περισσότεροι που πήγαν στη Συρία και το Ιράκ ε, προέρχονται από σημεία του Βελγίου όπου δραστηριοποιείται πολύ ιδιαίτερη οργάνωση αυτή, Σαριά for Belgium. Το δεύτερο κύμα όμως Βέλγων που έφυγε και πήγε εκεί βρέθηκαν μέσα από το διαδίκτυο. Ζητήθηκε από την πρώτη γενιά που γύρισε να βρούνε φίλους, συγγενείς κτλ. Και, και να τους ζεστικοποιήσουν. Σε κάποιες χώρες υπάρχει κάποια σταθεροποίηση, Βέλγιο, Ενωμένο Βασίλειο, στη Γαλλία ή στη Γερμανία δεν έχει σταματήσει. Οπότε θα έλεγα ότι δεν έχουμε καταφέρει να σταματήσουμε ούτε καν να περιορίσουμε τη ροή. Τέλος, θέλω να πω στον κύριο Μπασίρ για την έλλειψη χρηστής διακυβέρνησης. Συμφωνώ μαζί σας. Όντως θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει περισσότερα πράγματα μετά την Αραβική Άνοιξη. Θα έπρεπε όντω να ασχοληθούμε περισσότερο με τη μεταρρύθμιση στον τομέα τη ασφάλεια. Με την Τινησία, για παράδειγμα, συνεργάζομαι προκειμένου να του βοηθήσουμε να οικοδομήσουν εκ νέου την ασφάλεια στη χώρα του. Πρέπει να αρχίσουν από την αρχή οι υπηρεσίε ασφάλεια, να προωθήσουμε περισσότερο το κράτος δικαίου, να έχουμε ευφυεί πολιτικές για την πρόληψη. Ευτυχώς ο Πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος το θέλουν. και νομίζω ότι είμαστε σε θέση να βοηθήσουμε. Για άλλες χώρες, την για τη Λιβύη για παράδειγμα, επί του παρόντος δεν είναι δυνατόν. Θα είναι πολύ δύσκολο και τα επόμενα χρόνια. Άλλες χώρες όμως χρειάζονται περισσότερη στήριξη στον τομέα της ασφάλειας. Αυτά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η κυρία Φορτίγκα έχει κάτι να πει. Σύντομα παρακαλώ. Πολύ σύντομα. Κύριε Ντεκέρκοφ, η ερώτησή μου αφορά τη Ρωσία, Ιράν και Τουρκία. Αυτή την ερώτηση. Ας αφήσουμε την Τουρκία. Δεν απαντήθη. Δεν υπήρχε αίτημα για βαθύτερη συμμετοχή. Απλώς ρήτωση για το ποια είναι η κατάσταση. Άρα αυτό συνεπάγεται μια ανάγκη εμβάθυνσης των προσπαθειών. Έχετε κάποια σχόλια, λέει ο Πρόεδρος. Μπορείτε να αναλύσετε περισσότερο, διευκρινίσετε την ερώτηση για να απαντήσω. Τι εννοείτε ποια είναι η κατάσταση με το Ιράν και τη Ρωσία. Θα εξηγήσετε την ερώτησή σας. With Russia, very simply, I Απλώς με τη Ρωσία. Σας έδωσα ένα παράδειγμα. Το διάταγμα για την απαγόρευση διέλευσης από και προς το Αφγανιστάν. Όταν μιλάμε για συμμετοχή της Ρωσίας στα αντιτρομοκρατικά ε, μέτρα, αυτό ήταν που έκανε ήταν κάτι αντίθετο με τις προσδοκίες μας. Όσον αφορά το Ιράν, απλώς περιέργεια ήταν. Υπάρχει δυνατότητα το Ιράν να βοηθήσει για τη στήριξη μειονοτικών ομάδων όπως είναι οι χριστιανοί και οι γιαζίδοι, οι χαλδαίοι στο Ιράκ. Ήταν συγκεκριμένη ερώτηση. Εγώ δεν ασχολούμαι με το Ιράν. Σε αυτή τη φάση δύσκολο να σας απαντήσω αν μπορούμε να πετύχουμε κάτι με το Ιράν. Προσπαθούμε ο Πρωθυπουργό του Ιράκ να έχει μια πιο ολιστική πολιτική. Ό,τι πετύχουμε εκεί είναι καλό. Για τις πυρηνικές διαπραγματεύσεις δεν συμμετέχω τόσο πολύ να πω ότι γίνονται τέτοιες συζητήσεις στο περιθώριο των διαπραγματεύσεων. Η ύψιστη προτεραιότητα είναι αυτή των διαπραγματεύσεων. Τα πυρηνικά εννοεί. Και χρειάζεται τον περισσότερο χρόνο. Εξέφρασα προσωπικές απόψεις. Είπα όταν αυτό διευθετηθεί, με τα πυρηνικά δηλαδή, θα πάμε και στα άλλα. Ε, καλή ιδέα αυτή η δική σας. Για τη Ρωσία κάτι άλλαξαν βοηθάει ο Πρόεδρος να εξηγήσει στον κύριο Ντεκέρκοφ την ερώτηση. Α, Ρωσία. Όλες οι συζητήσεις που είχα με τους ομολόγους μου, τους Ρώσους, είναι μέλη του φορέα του GTCF όπου συζητάμε και αυτοί ανησυχούν για τις εξελίξεις όσον αφορά το Ισλαμικό κράτος, τον Daesh Πρέπει να βαθυθεί οι σχέσεις μας. Δεν είναι τόσο εύκολο τώρα όσο ήταν παλιά, πριν την κρίση στην Ουκρανία. Αυτό είπα λοιπόν. Για την αξιολόγηση σε μεγάλο βαθμό έχουμε και εμείς τις ίδιες ανησυχίες όσον αφορά τον Ντάις και την Αλκάιντα. Οι απόψεις για το Αφγανιστάν επίσης ε, πλησιάζουν. Ευχαριστώ πολύ κύριε Ντεγκέρχοφ, λέει ο κύριος Πάσκου. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα άλλο βήμα στο διάλογό μας. Ευχαριστώ που ήρθατε. Θα τα ξαναπούμε την επόμενη φορά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας εύχομαι ό,τι καλύτερο. Θα ήθελα να κοινώσω στους συναδέλφους ότι το επόμενο σημείο επίσκεψη στην Τεχεράνη που θα παρουσιαστεί από τον πρόεδρό μας τον κύριο Μπροκ διεξάγεται και κλεισμένον των θυρών η συζήτηση αυτή.